Okay, ladies Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως. Λοιπόν, αγαπητοί συναδελφοί, συνεχίζουμε τη συνεδρίαση. Περνάμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Η παρουσίαση και συζήτηση με τον πρέσβη μας για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τον κύριο Πανγκράτ. τον οποίο καλωσορίζω θερμά. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου συχνά είναι στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Ιδίως μετά την επίτευξη παρά τα άσχημα προγνωστικά κάποιων επιτυχιών στο Μπαλί και ε, αναμένεται να υπάρξουν και άλλα βήματα εντός του ΠΟΕ, ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν. Αυτή η ελπίδα όμως δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής. Απέτυχαν ε, οι προσπάθειες για να υπάρξει συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου. Γιατί φαίνεται ότι τα εμπόδια είναι μεγαλύτερα από ό,τι θεωρείται. Έτσι έχει η κατάσταση. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΠΟΕΜ και το Φεβρουάριο την ε, Υπουργική Συνέλευση. Οπότε νομίζω ότι είναι σκόπιμο τώρα να σκεφτούμε πώς θα πρέπει να λειτουργήσει ο ΠΟΕΜ και πώς θα τον αντιμετωπίσουμε περαιτέρω. Κύριε Πρέσβη, το ερώτημα που τίθεται πάντα είναι, είναι σκόπιμο να υπάρχει αυτός ο ΠΟΕ ή πιο χρήσιμες είναι τελικά οι διμερείς επαφές και διακανονισμοί. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Και η συζήτηση πέρα από τις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις σχετίζεται και με άλλα ζητήματα και είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη του ΠΟΕ. Είναι ένα θέμα που τίθεται συνολικά από την ε, πολιτική ηγεσία που θέλει να ε, προωθήσει την πολυεθνική αντιμετώπιση. Πολλές ερωτήσεις λοιπόν. Κύριε Παγκράτη, χαίρομαι για την παρουσία σας. Σας καλωσορίζω, έχετε το λόγο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι πολύ ευτυχής που μου δίνετε αυτή η ευκαιρία να απευθυνθώ σε εσά και να σας μιλήσω για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ε, θα αναφερθώ σύντομα στην σημασία του, ε, των ε, πολυμερών διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ και ε, θα εξειδικεύσω για την ε, κατάσταση στην οποία βρίσκονται ε, οι συμφωνίες διευκόλυνσης καθώς επίσης και η συμφωνία Μπαλή και μετά Μπαλή. Και βεβαίως θα αναφερθώ και με γενικότερους όρους για στην παρούσα κρίση που διανύει ο οργανισμός που ενδεχομένως δεν θα είναι μία από τις πολλές κρίσεις αλλά ενδεχομένως αυτή η μία κρίση η οποία θα οδηγήσει σε βαθιές αλλαγές στις διαπραγματευτικές αρχές και διαδικασίες θα επικεντρωθώ κυρίως σε προβλήματα και προκλήσεις και δυσκολίες των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην λησμονούμε το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει η χώρα η συζήτηση αυτή. Ο ΠΟΕ είναι ε, κάτι περισσότερο από διαπραγματευτικό ε, σώμα. Έχει και άλλες λειτουργίες. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, ασχολείται επίσης με επίλυση διαφορών. Αυτό είναι κάτι μοναδικό μοναδικό και δεν υπάρχει, ε, δεν υφίσταται κάτι ε, αντίστοιχο σε άλλες ε, περιπτώσεις ε, και έστω και αν έχουν γίνει προσπάθειες να οικοδομηθεί κάτι αντίστοιχο. Επίσης δεν υπάρχει τίποτα συγκρίσιμο όσον αφορά ε, τις, τους παγκόσμιους οργανισμούς. Επίσης έχει την λειτουργία της επιθεώρησης και επιτήρησης που είναι πάρα πολύ σημαντικός ρόλος ειδικά όσον αφορά την αποτροπή των κρίσεων ε, που μπορούν να προκληθούν λόγω κάποιου βαθμού προστατευτισμού. Επίσης, πολύ συχνά υπάρχει και αυτή η λεγόμενη συνήθις εργασία που συχνά ε, υποτιμάται, δηλαδή η διαχείριση και η υλοποίηση υφισταμένων ε, συμφωνιών. Και στον τομέα αυτό η διάσταση της αποτροπής ή της επίλυσης τρυφών και διαφωνιών είναι μια πάρα πολύ σημαντική λειτουργία. Υπάρχουν και άλλες λειτουργίες οι οποίες είναι επιχειρησιακές και οι οποίες λειτουργούν ανεξάρτητα από τις διαπραγματευτικές ε, λειτουργίες. Ωστόσο, ε, αποδυναμούμενη η διαπραγματευτική δυνατότητα ε, αποδυναμούνται και ολόκληρη, όλες οι άλλες διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στον ΠΟΕ. Ε, και βεβαίως οι δυσκολίες απεικονίζονται ε, και από το γεγονός ότι έχει 160 μέλη, 23 χώρες ε, ήδη έχουν υποβάλει αίτηση και βρίσκονται σε διαδικασία αποδοχής της υποψηφιότητάς τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά και ορισμένα εξειδικευμένα πλεονεκτήματα. Θα αναφερθώ σε ορισμένα εξ αυτών πολλά από τα κεντρικά στοιχεία της διεθνούς διαπραγμάτευσης όπως ας πούμε ε, επίλυση ε, τριβών και διαμαχών οι οποίες ε, σχετίζονται με εσωτερικές επιδοτήσεις και αγροτικές επιδοτήσεις κτλ. Εδώ υπάρχει ένα πλεονέκτημα στην επίλυση αυτών επίσης. Αναγνωρίζεται ότι οι διεθνείς, οι διμερείς, συγγνώμη, συμφωνίες μπορούν να προκαλέσουν έναν κατακαιρματισμό όσον αφορά τις νομοθετικές και λοιπές ρυθμίσεις. Άρα ε, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των προβλημάτων ε, για τις εμπορευόμενες επιχειρήσεις ε, και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εμείς μπορούμε μέσα σε πλαίσια πολυμερών διαπραγματεύσεων να εξειδικεύσουμε σε, λαμβάνοντας υπόψη τις διμερείς συμφωνίες. Επίσης, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ε, είναι, ε, λαμβάνουν χώρα ε, οι συζητήσεις με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί δηλαδή αποκτούν φωνή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να λησμονούμε επίσης κάτι προφανές, δηλαδή ότι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να ονομαστεί πολύ διμερές ε, παράδοξο όπου δηλαδή ε, όπου αυξάνεται η αλληλεξάρτηση και επομένως χρειαζόμαστε περισσότερες κοινέ λύσεις. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα πρέπει να πω ότι είμαστε όλο και σε πιο δυσχερή θέση. Δεν είμαστε σε θέση δηλαδή να, ε, ε, να, να ολοκληρώσουμε ε, διαδικασίες. Βεβαίως υπάρχουν προτεραιότητες με την έννοια βεβαίως ότι είμαστε πάντα απολύτως δεσμευμένοι, απολύτως στρατευμένοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι ώστε ε, να ε, προετοιμάσουμε ε, τις ε, πολυμερείς συμφωνίες και βεβαίως και σαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς στη Γενέβη είμαστε πάντα έτοιμοι και προσπαθούμε να αποτρέψουμε καταστάσεις ή τέλος πάντων να, έχουμε, να αναλάβουμε δράσεις πριν να εμφανιστούν τα προβλήματα. Βεβαίως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου όπως είπατε και εσείς είναι μοναδικός αλλά γιατί Ακριβώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει μοναδικό ρόλο ε, στα πλαίσια ε, του ε, ΠΟΕ και φυσικά στις γενικές εξωτερικές μας σχέσεις είναι το χώρος στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάντα μία φωνή την οποία εκφράζει μέσα από έναν ενιαίο μοναδικό διάβλο τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν ε, ότι ε, ε, οι θέσεις είναι διεθνούς ενδιαφέροντος, είναι μεγάλη επιρροή μας και επομένως μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας. Επίσης υπάρχει μια διαμεθοραϊκή αναγνώριση του ΠΟΕ ως μεγάλη δύναμη και ως ε, δυνάμενος να ε, βρει συμβιβαστικές λύσεις. Επιτρέψτε μου επίσης κύριε Πρόεδρε να πω ότι έχοντας ε, η 30 ετή εμπειρία σε διεθνές εμπόριο πρέπει να ομολογήσω ότι είναι μοναδική εμπειρία μου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου γιατί μπορεί να αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και επιρροή. Τώρα να περάσουμε στις διαπραγματεύσει, γιατί αυτό θέλετε να ακούσετε. Τα στοιχεία είναι καθαρά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δημιουργήθηκε το 1995, ε, ενώ το DDA ξεκίνησε το 2001 ε, ε, και ε, πρόκειται για απάβγασμα κατά κάποιο τρόπο των προσπαθειών που είχαν καταβλήθει μέχρι τότε και 7 μήνες μετά από την συμφωνία του Μπαλί η οποία δυσκολεύτηκε γιατί υπήρχε μία χώρα η οποία δεν συμφωνούσε με ένα στοιχείο από, την, τα όσα συμφωνήθηκαν στο Μπαλί. Πρέπει να πούμε ότι μέσω της κατάστασης αυτής το ε, βλέπει ότι δυσκολεύεται τελικά να υλοποιήσει τις, ε, τις ε, αποφάσεις και τελικά βλέπουμε ότι καταλήγουμε σε κείμενα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις ούτε δίνονται να χρησιμοποιηθούν και ούτε χρησιμοποιούνται τελικά. Ε, εμείς θέλουμε ένα, να αλλάξουν τα πράγματα γιατί πραγματικά ε, ε, ελοχεύει ο κίνδυνος ο οργανισμός να γίνει ένας οργανισμός κατά κάποιο τρόπο παγωμένος ο οποίος δεν βρίσκεται σε νάρκη πούμε και δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Πιστεύουμε ότι μέσω των αποτελεσμάτων του Μπαλί μπορούμε να αφυπνιστούμε και μπορούμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να βρούμε τρόπο ε, ε, ένας ενδιαφέρον και σημαντικός παγκόσμιος οργανισμός να βρει τον τρόπο να προσαρμοστεί στις νέες ε, συνθήκες. Βεβαίως θα πρέπει να λειτουργήσουμε σωστά έτσι ώστε αυτή η δύσκολη μεταβατική περίοδος η οποία ξεκίνησε το 2011 να ολοκληρωθεί σωστά. Αποφασιστικό ρόλο θα παίξουν οι επόμενες εβδομάδες και θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω τι εννοώ. η διαδικασία που ξεκίνησε το 2011 ε, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ε, ε, ξεκίνησε ακριβώς γιατί καταλάβαμε ότι είχαμε προβλήματα όσον αφορά την υλοποίηση των συζητήσεων και των αποφάσεων. Και ξεκίνησε λοιπόν αυτή η διαδικασία αμφισβήτησης και αλλαγής. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα είχε πάρα πολύ περιορισμένο περιοριστική εντολή και επομένως δεν είχε ένα περιθώριο ελιγμών. Ταυτόχρονα όμως ε, αυτό το ε, κανονιστικό πλαίσιο το οποίο ήταν σφιχτό ε, ήταν, έφτασε να είναι υπερβολικά σφιχτό και περιοριστικό και επομένως όλη αυτή η διαδικασία κατέληγε τελικά σε μια δημιουργία εγγράφων τα οποία δεν είχαν καμία ουσία και σημασία. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε ε, να ε, ε, προσθεθεί ευελιξία έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με πιο ευέλικτο τρόπο και επομένως να διερευνηθούν νέοι καινοτόμοι τρόποι διαπραγμάτευσης και συμφωνίας. Θα πω εξ αρχής ότι δεν υπήρξαν αλλαγές στο πνεύμα των κειμένων ε, επί των οποίων είχε βασιστεί η ε, δράση μας, αλλά ε, μία κοινή διαπίστωση ότι κάποια πράγματα έπρεπε να αλλάξουν ε, και βεβαίως ε, η δυνατότητα πλέον ε, κατέστη φέσο ότι η δυνατότητα να βρεθούν συμφωνίες μεταξύ τόσων πολλών χωρών δημιουργούσε πολλά προβλήματα τα οποία οδήγησαν στην βαθιά κρίση και η οποία με τη σειρά της οδήγησε στην ανάγκη αλλαγών. Έγινε λοιπόν, ε, ξεκίνησε λοιπόν μια προσπάθεια έτσι ώστε να βγούμε από αυτά τα στενά χαρακόμματα και να μπορέσουμε ε, να ε, ξεπαγώσουμε τον οργανισμό πρέπει να σας πω ότι το 2011 υπήρξε ένας κύριος ε, παράγων, ε, δηλαδή ε, γιατί είχε αλλάξει πλέον ο κόσμος σε σχέση με την εποχή κατά την οποία είχε οριστεί η εντολή. Εν τω μεταξύ είχαν αναπτυχθεί οι αναπτυσσόμενες χώρες, υπήρξαν οι αναδυόμενες οικονομίες οι οποίες άλλαξαν την αρχιτεκτονική και η πρόσβαση στην αγορά είχε πλέον αλλάξει εντελώς. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, δυσκολίες ε, και φυσικά ε, εάν προχωρήσουμε και κάνουμε όλες τις διαδικασίες έτσι ώστε να κάνουμε τις σημαντικές αλλαγές τότε θα αντιμετωπίσουμε ακόμα περισσότερες δυσκολίες αλλά ωστόσο πρέπει να βλέπουμε λίγο και γύρω μας. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, ο κόσμος έχει, γίνει, έχει αλλάξει και έχει γίνει πολύ πιο περίπλοκος και επομένως δεν μπορεί ο ΠΟΕ να παραμείνει στάσιμος. Το Μπαλί ακριβώς κατέδειξε την περιπλοκότητα του κόσμου στην οποία καλείται τρόπο λειτουργήσει. Ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες αυτές, αλλά παραμένοντας με τα πόδια στη γη, παραμένοντας ρεαλιστές. Ε, επομένως, ε, ξεκίνησε αυτή η μεγαλύτερη ευελιξία από το MCA του 2011 και συνεχίστηκε και στον Παλί βρήκαμε ένα νέο τρόπο ε, να, δημιουργούμε το, ε, το θεματολόγιό μας, την ατζέντα μας ε, και ένα νέο τρόπο προσέγγισης των προβλημάτων από κάτω προς τα πάνω. Βασιστήκαμε σε ζητήματα τα οποία ενδιαφέρουν όλους. Ας πούμε, η διευκόλυνση του εμπορίου είναι κάτι διατομεακό και είναι κάτι το οποίο αφορά και ενδιαφέρει όλες τις χώρες. Ε, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ε, μία ε, άλλη ισορροπημένη διαδικασία η οποία βασίστηκε στις 10 αποφάσεις του Μπαλί. Επομένως, μία νέα είπαμε ισορροπία ε, μέσω της οποίας μπορούμε να φτάσουμε σε συγκλήσεις. Θα ήθελα να επιμείνω στο ότι το Μπαλί δεν ήταν μια συγκυρία και δεν έτυχε απλώς. Αποτέλεσε το επιστέγασμα πολλών προσπαθειών και μάλιστα στοχευμένων προσπαθειών ε, ήταν επίσης αποτέλεσμα της ευελιξίας ε, η οποία ε, προστέθηκε στα κείμενα και η οποία έδωσε την δυνατότητα να φτάσουμε ε, και βεβαίως υπήρξαν και άλλοι παράγοντες όπως ας πούμε οι θεωρήσεις όπως είναι ε, τροφιμικά, μη τροφιμικά, περιβαλλοντικά ζητήματα ε, τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ και συνέβαλαν στην αλλαγή κλίματος στις διαπραγματεύσεις στη Γενέβη. Είμαι απολύτως πεπισμένος όπως και όλοι μας στη Γενέβη ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τις πολυμερείς συμφωνίες εάν και με την προϋπόθεση ότι όλοι θα καταβάλουν καταβάλουν τις ίδιες προσπάθειες με την προϋπόθεση ότι ε, θα αποκομίσουμε τη σοφία των παρελθόντων ε, ετών και ε, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να δώσουμε αυτό το μεγάλο βήμα προς τα εμπρός έτσι ώστε να γίνει αυτή η μεταμόρφωση. Βεβαίως η μεταμόρφωση δεν είναι μοναδική, έχει και, άλλες, άλλα στοιχεία. Τώρα με τη νέα κρίση ήταν προφανές την τελευταία μέρα των διαπραγματεύσεων στον Παλί, ιδιαίτερα την τελευταία μακρά νύχτα μέχρι τα ξημερώματα, οπότε και καταλήξαμε, ήταν σαφές αυτό που αποκαλώ η αρνητική δύναμη του ενός, εφόσον χρειάζεται ομοφωνία. Όσο θαυμάσια και είναι η διαδικασία με βάση ωραία θέματα και υπάρχουν συγκλήσεις, διαπραγματεύεσαι ένα αποτέλεσμα που το αποδέχονται όλοι, αλλά αρκεί μόνο ένα μέλος που είναι αποφασισμένο να πάει προς άλλη κατεύθυνση ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά τη συμφωνία, για να μπλοκάρει την όλη διαδικασία. Και αυτό είναι βεβαίως ανησυχητικό και για το μέλλον. Και δεν λέω ότι πάντα είναι ο ίδιος που ε, ασκεί βέτο. Θεωρώ λοιπόν ότι και στο μέλλον, εάν συνεχίσουμε να διαγματευόμεθα και περάσουμε σε πιο σημαντικά θέματα, θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος βέτο. Ποια είναι τώρα η κατάσταση. Πολύ δύσκολη. Πολύ σοβαρή, όπως είπε και ο Ζαν Λουκ Ντεμαρτή σήμερα το πρωί. Εάν ένα μέλος αρνηθεί να εφαρμόσει ένα σημαντικό τμήμα του πακέτου του Μπαλί, για παράδειγμα, υποχρέωση να υπογραφεί το πρωτόκολλο για την διευκόλυνση εμπορίου μέχρι 31 εβδόμου. Είναι σαφής αυτή η εντολή, δεν είναι να γίνει κάποια διαπραγμάτευση σε κάποια φάση, να καταλήξουμε κάπου. Ήταν δέσμευση να εφαρμοστεί κάτι μετά από την νομική βέβαια επαλήθευση. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν το έπραξαν όλοι αυτό, ένα συγκεκριμένος, τουλάχιστον ένα μέλος δεν το έπραξε, σημαίνει ότι δεν ε, λειτουργεί το σύστημα. Δεν μπορούμε να το αναδιαπραγματευτούμε. Δεν είναι εύκολο να επαναληφθεί μια τόσο περίπλοκη διαδικασία. Μια τόσο μακρόχρονη διαδικασία προσπάθειας εξισορρόπησης συμφερόντων που αντανακλάται σε 10 αποφάσεις άμα του βγάλεις ένα κομμάτι, ένα συστατικό, να επιχειρήσεις να, να τα υπόλοιπα, είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι ότι κάποιος δεν θέλει. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο για την οργάνωση. Αν αποδεχθούμε κάτι τέτοιο, τότε και άλλοι θα επανέλθουν επί άλλων θεμάτων της συμφωνίας. Δεν μπορούμε να ξαναδιαπραγματευτούμε τον παλί. Ούτε και την μετάμπαλή κατάσταση. Για τους ίδιους λόγους. Δεν υπάρχει συμπεφωνημένη βάση επί της οποίας να διαπραγματευτούμε την μετά μπαλή κατάσταση. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι πολύ απαιτητικό, πολύ δυσχερές να δούμε πώς. Αλλά αυτή η δυσχερής κατάσταση στην οποία ε, βρισκόμαστε δεν οφείλεται στην ουσία των ετοιμάτων που μας υποβάλλονται αλλά η δυσκολία είναι η σύνδεση μεταξύ της ε, διευκόλυνσης εμπορίου και το σύστημα ε, δημόσιας συσσόρευσης που έχει η Ινδία. Είναι θέμα επιστημιστικής ασφάλειας για αυτούς και πολύ ευαίσθητο εσωτερικά. Η επιστημιστική ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό θέμα για όλους μας. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Ίσως είναι σύστημα αποθήκευσης περισσότερο τροφίμων. Ε, οπότε, επειδή έχουμε και μία ρήτρα ειρήνης για κάποιες πρακτικές ε, της Ινδίας και άλλων αναπτυσσόμενων χωρών για τη δημόσια αποθήκευση. Είπαμε ότι έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν τις πρακτικές μέχρι να υπάρξει μόνιμη λύση. Και θέλουμε βεβαίω να επιταχυνθεί η εξέβρεση λύση. Είπαμε στον Παλίο ότι θα βρούμε μόνιμη λύση μέχρι το 2017. Τώρα η Ινδία ε, θέλει να υπάρξει πιο σύντομα λύση. Σημαντική αυτή η απέτηση. Και για άλλα αναπτυξιακά θέματα ε, έχουν, γίνει, ε, έχουν υποβληθεί αιτήματα να βρούμε πιο σύντομα λύση. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Κανείς μεταξύ των κρατών μελών δεν είναι κάθετα εναντίον αυτών των ετοιμάτων. Όμως η πραγματική δυσχέρεια είναι αυτή η σύνδεση με την διευκόλυνση του εμπορίου και το μπλοκάρισμα του πρωτοκόλου διευκόλυνσης εμπορίου. Γιατί δεν σέβεται τον παλί. Δεν, σέβεται, δεν σέβονται τέτοια αιτήματα την συμφωνημένη βάση. Είναι κάτι, ένα θέμα τακτικής, είναι πολιτικό θέμα αυτό. Δεν είναι επί της ουσίας είναι αυτή η προσπάθεια τακτικής για πολιτικούς λόγους υποβάλλονται αυτά τα αιτήματα και δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε. Είμαστε λοιπόν σε πολύ επικίνδυνη θέση λόγω αυτής της σύνδεσης των θεμάτων. Πολλά μπορούμε να πούμε για διάφορες πλευρές, αλλά αυτό είναι ο ουσιώδης κίνδυνο. Αυτή η σύνδεση που γίνεται μεταξύ αυτών των θεμάτων. Μου θυμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε με τα δάση των χωρών της Μεσογείου. Όταν υπάρχει μία πυρκαγιά των δασών μπορεί να αναγεννηθεί. Εάν καεί και δεν παρεύεις μετά, ξαναγίνεται. Μπορεί να ξαναγίνει εκατοντάδες φορές. Αλλά υπάρχει μια κρίσιμη στιγμή αν κάψει ένα δάσο και βγουν τα καινούρια δέντρα, τα νέα δέντρα και τη στιγμή που φτάνουν σε κάποιο ύψο, ξανακαούν τότε έχουμε χάσει τους ε, παλιούς σπόρους ενώ δεν έχουν παραχθεί νέοι και το δάσος δεν μπορεί να αναγεννηθεί πλέον. Ο ΠΟΕ, ξέρετε, πολλές φορές έχει αναγεννηθεί στη φάση διαπραγματεύσεων, αλλά τώρα είμαστε σε επικίνδυνη φάση. Είναι αυτός ο συνδυασμός έλλειψη σεβασμού των δεσμεύσεών μας σε μια κρίσιμη στιγμή που μόλις είχε αρχίσει να επανακτά αξιοπιστία ο οργανισμός. Λόγω της κατάστασης αυτής και καταλήγω, καταλήγω στα εξής σημεία. Τι θα γίνει στο μέλλον από εδώ και πέρα. Η πολυμερής ε, μέθοδος, ε, την οποία ε, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε από 31η Εβδόμου, λόγω της κατάστασης που ελπίζω σαφώς να σας εξήγησα. Μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτήν. Πρέπει να αφήσουμε επαρκές χρονικό διάστημα και επί της ουσίας κάποια περιθώρια στην Ινδία και άλλες χώρες για να επανέλθουμε στην πολυμερή διαδικασία. Εφόσον βεβαίως επανέλθουμε στα πλαίσια των, διαδικασιών, των αποφάσεων του Μπαλί. Βεβαίως συζητήσεις αλλά σεβόμενοι αποφάσεις του Μπαλί. Αυτή είναι η κύρια προτεραιότητά μας. Αυτή θα ήταν η βέλτιστη λύση. Τώρα μη μου ζητήσετε να σας πω τι ποσοστό επιτυχίας ε, έχει, θα έλεγα όμως ότι είναι μη μηδενικό. Αλλά εάν παρακολουθήσει κανείς την ε, εσωτερική πολιτική της Ινδίας, σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο. Πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να επανέλθουμε στην πολυμερή προσέγγιση. Δεύτερον, εάν το τρέχον αδιέξοδο συνεχιστεί μερικές ακόμη εβδομάδες, γιατί δυστυχώ ο χρόνος είναι εναντίον μας, η κρίση που θα προκύψει θα είναι η χειρότερη στην ιστορία του ΠΟΕ. Τρίτον, αν συμβεί αυτό, πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας, όταν θα εξετάσουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον, ότι η χειρότερη περίπτωση για την Ένωση και την μεγάλη πλειονότητα των μελών της και των μελών του ΠΟΕ θα είναι ότι η κρίση θα ξαναπαγώσει τον ΠΟΕ. Το πακέτο του Μπαλί και η διευκόλυνση εμπορίου θα χαθούν. Κανένα δεν συμφέρει αυτό. Τέταρτον, όπως είπα και προηγουμένως, εξήγησα ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε τις θέσεις των μελών το Μπαλί έδωσε την εντύπωση στα περισσότερα μέλη στη Γενέβη ότι μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Και όλοι θέλαμε να μην χάσουμε τα κεκτημένα του Μπαλί. Και λοιπόν τη συμφωνία για διευκόλυνση εμπορίου. Οι περισσότερε αναπτυσσόμενες χώρε θέλουν τη συμφωνία αυτή και όλα τα συμπαραμαρτούντα. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη υπάρχουν ήδη άρθρα και Θα αρχίσουν να εξετάζουν το ενδεχόμενο πολυμερών εναλλακτικών λύσεων αν επιβεβαιωθεί η προθεσμία. Και μπορεί να γίνει υποχρεωτική αυτή η προσέγγιση αν οι πολυμερει ε, επιλογέ είναι οι μόνε που θα απομένουν ανοιχτέ. Πέμπτον, σε μια τέτοια περίπτωση θα έχουμε δυσχέρειε. Ο ΠΟΕ θα βυθιστεί σε μια κρίση που μπορεί βέβαια να οδηγήσει σε πολλέ ε, αλλαγέ του θα ξεκινήσουμε μια θεμελιώδη συζήτηση για το μελλοντικό του ρόλο και τις μελλοντικέ μεθόδους εργασίας. Και έκτο, εάν γίνει κάτι τέτοιο, η Ένωση θα ακολουθήσει πάντα τις αρχές που έχουμε ακολουθήσει στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις. Ότι θέλουμε η λύση να μείνει εντός του ΠΟΕ, να ευνοήσουμε πολυμερεί λύσεις, σε κάθε δυνατό βαθμό θα επιδιώξουμε πάντα την πολυμεροποίηση. Εστιάζοντας λοιπόν σε πολυμερείς επιλογές, ούτω ώστε τον παλί να οδηγήσει στο DTA και να επιτρέψει στον, λειτουργό, στον οργανισμό να λειτουργήσει στον 21ο αιώνα. Αυτά νομίζω είναι. Αυτές είναι οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές μας. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι να αποφύγουμε το χειρότερο σενάριο, η οργάνωση δηλαδή, να παγώσει εκ νέου. Πρόεδρε, τελείωσα. Μάλλον τελειώνω, τονίζοντας ότι η Ένωση παίζει τα τελευταία χρόνια κύριο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια τη μεταβατική. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε αυτό τον ρόλο και έχουμε την πρόθεση. Η συμβολή της Επιτροπής σας θα είναι ουσιώδης σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να συνοψίσω την κατάσταση όπως την θεωρώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Θαυμάσια, κύριε Πρέσβη. Σας θαυμάζω για το πνεύμα αισιοδοξία που φέρατε στην αίθουσα. Αυτό είναι δύσκολο, αν έχει κανείς υπόψη πολλά όσα λέγονται για τον ΠΟΕ. Ξέρετε θαυμάσια βεβαίως ε, την, ε, τον ΠΟΕ. Πραγματικά σας συγχαίρω για όσα μας είπατε. Τώρα θα πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι. Πρώτα η κυρία Μακλάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρέσβη για τις απόψεις σας έτσι όπως τις εκφράσατε σήμερα. Νομίζω ότι το μότο σας είναι το ίδιο, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον. Και εγώ το ίδιο έχω. Ε, παρακολουθώ πιο στενά τώρα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ε, και στο τέλος της, ε, ε, του διορισμού σας ε, θεωρείτε ποια θεωρείτε ότι θα είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα και στα πλαίσια του μότο τίποτα δεν είναι, της αρχής τίποτα δεν είναι αδύνατο. Τι πιστεύετε όσον αφορά τον κανόνα της ομοφωνίας στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας αλλαγής, πορείας και δυνατότητας λήψης αποφάσεων. Τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Judith. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση που μας κάνατε όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Ε, λέτε ότι εάν δεν ε, κινηθούμε στα πλαίσια του ΠΟΕ θα δούμε πληθώρα ε, διμερών ε, συμφωνίων, αλλά το βλέπουμε ήδη. Πρόκειται για συμφωνίες οι οποίες γίνονται παράλληλα με τις συμφωνίες και τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ. 18 μήνες ε, μετά από την ε, συνθήκη βλέπουμε ότι του Μπαλί βλέπουμε ότι είναι λίγες και ούτως ή άλλως μεγάλη συζήτηση γίνεται ε, γιατί οι χώρες BRICS δεν έχουν συμμετάσχει στις ε, διαπραγματεύσεις. Ε, ποιες είναι, ποια είναι η άποψή σας επίσης σε σχέση με την Ουρουγουάη και την Κίνα και τις υποψηφιότητες τους. Επίσης ενδιαφέρον θα ήταν να μας πείτε την άποψή σας για τον τρόπο με τον οποίο προχωρούν οι διαπραγματεύσεις γιατί ο πω είναι μέρος ανεπίσημο στις διαπραγματεύσεις αυτές. Βλέπετε να επιτευχθεί η κριτική μάζα Thank you. για τη συμφωνία αυτή για το εμπόριο και τις υπηρεσίες. a lot. I mean... Ευχαριστώ. Ε, πάλι για αυτή τη συμφωνία για την ΤΙΣΑ. ποιος είναι ο και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος ε, της, του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ε, σε ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να ε, προχωρήσει ε, βεβαίω ε, μα το είπατε κι εσείς ότι πάντα είχε δημιουργήσει συμφωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίω ακούμε πολλά, βλέπουμε πολλά αλλά ε, επί του πρακτέου τα πράγματα είναι διαφορετικά και έχω την αίσθηση και φαντάζομαι ότι δεν είμαι η μόνη ότι οπωσδήποτε έχει χαθεί το ενδιαφέρον για την πολυμερότητα για κάθε είδους ε, συμφωνίες. Κοιτάξτε, εσείς ε, ε, έχετε την έδρα σας στην Γενέβη, τα βλέπετε όλα από κοντά. Ποια είναι η προσωπική σας εμπειρία για το πόσο θα αξιολογηθεί αυτή η εργασία που γίνεται στη Γενέβη εξακολουθεί να είναι το κέντρο ή μήπως τα τελευταία χρόνια έχει λίγο αλλάξει αυτό το κέντρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι πριν τον Παλί έβλεπα τα πράγματα διαφορετικά. Τώρα μπορώ μετά τον Παλί να συμμεριστώ την αισιοδοξία σας. Αναφερθήκατε και λίγο στην πολιτική κατάσταση στην ε, Ινδία. Βλέπετε να υπάρχουν δυσκολίες και σε άλλες χώρες εκτός από την ε, ε, Ινδία. Ε, υπάρχει επίσης σε περίπτωση που αυτός ο φραγμός, α πούμε η δυσκολία της Ινδίας εξεκολουθεί, υπάρχει ένα, μια εναλλακτική λύση, ένα εναλλακτικό ε, σενάριο ή ε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, καμία εναλλακτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που ξανά ήρθατε στην Επιτροπή μας. Μας εξηγήσατε την ε, κατάσταση ε, και, τις, ε, και λέτε ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης επί της ουσίας. Ναι, βεβαίως πάντα υπάρχει είτε η ευκαιρία είτε ο κίνδυνος να πάει κανείς προς τα πίσω, γιατί ε, υπάρχει έτσι κι αλλιώς και ο, ο σκληρός νόμος και ο ήπιος νόμος hard law και που είναι αυτός του εμπορίου, που είναι αυτός των ε, οικονομιών που ηγούνται κτλ. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει soft law, ε, οι προσπάθειες δηλαδή να ε, φτάσουν σε αυτό το hard law και οι αναπτυσσόμενες χώρες. Και βεβαίως προκύπτει το ερώτημα και συμφωνώ μαζί σας το ζήτημα μάλλον ότι θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε επιστοδρόμηση. Ε, αλλά ε, πρέπει να καταλάβουμε πώς, ε, ποια είναι η πραγματικότητα στις χώρες αυτές, στην Ινδία και στο Πακιστάν. Αυτό το 10% ας πούμε της γεωργικής παραγωγής και το κατά πόσον θα μπορέσουν να φτάσουν στο ποσοστό αυτό. Αυτό θα σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ πιο ακριβά τα τρόφιμα, έστω και αν επιτευχθεί η συμφωνία και επομένως πώς η κυβέρνηση της Ινδίας πρέπει ή μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση ε, λαμβάνοντας υπόψη κιόλας ε, ότι ε, έγινε προσπάθεια αποφυγής πολιτικών συγκρούσεων στη χώρα αυτή και ήταν άλλωστε και το διακύβημα των εκλογών. Και η τωρινή κυβέρνηση στην Ινδία αντιμετωπίζει τα ίδια που είχε αντιμετωπίσει και η προηγούμενη. Ε, δεύτερο από τα έξι σημεία ήταν ο εκδημοκρατισμός της διαδικασίας ε, λήψης αποφάσεων στο Παγκόσμιο Οργανισμό ε, Εμπορίου. Πώς θα το κάνετε αυτό. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ακόμη έξι έχω ζητήσει το λόγο, οπότε θα κλείσω πλέον τον κατάλογο μιλητών. Ο Λόρδος Ντάτμουθ λοιπόν. Πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά θα περιοριστώ σε μια τεχνική ερώτηση ή δύο-τρεις. Οι εμπορικές συμφωνίες έχουν ε, αποκλειστικά, είναι αποκλειστικά ενωσιακή αρμοδιότητα από πριν από τη Συνθήκη και η χώρα μου δεσμεύεται από τις συμφωνίες αυτές από το 1975. Η κυρία Κέλλερ μίλησε για την εμπορική πολιτική της Ένωσης. Υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, τα μεμονωμένα κράτη-μέλη είναι μέλη του ΠΟΕ. Η Βρετανική κυβέρνηση, που γνωρίζω πώς λειτουργεί, στέλνει λοιπόν κάποιους εκπροσώπους, αλλά η έδρα, οι δυνατότητες δεν χρησιμοποιούνται. Ως πρέσβης στον ΠΟΕ της Ένωσης, πώς ε, συνεργάζεστε με τα κράτη-μέλη που έχουν ε, έδρες που είναι μέλη του ΠΟΕ, που στέλνουν εκπροσώπους. Επικρατεί πάντα η δική σας άποψη. Τους λέτε ορίστε αυτό είναι και να το έχετε υπόψη σας. Ή έρχονται και σας λένε ανησυχούμε γι' αυτό, α, για τα αυγά σε σκόνη για παράδειγμα. Μπορείτε να το κάνετε. Πώς λειτουργεί. Και μια που έχουμε το προνόμιο της παρουσίας σας, παρακαλώ εξηγήστε μας πώς γίνονται αυτά. Η κυρία Μόσκα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τρία γρήγορα ερωτήματα χρονικά. Το πρωί με την διαπόψεων. είπατε εσείς ότι πρόκειται για σύντομα χρονικά διαστήματα, δύο-τρεις εβδομάδες μόνο. Πέστε μου σας παρακαλώ, πώς έχει χρονικά το πράγμα για να δούμε για την επίλυση αυτών που είπατε, τι αποτέλεσμα θα μπορούσαμε να έχουμε. Κάτι ακόμα. Σήμερα το πρωί εσείς και πάλι τονίσατε κάτι ότι έχουν τεράστια σημασία οι χώρες και με, θα με ενδιαφέρε και εμένα να καταλάβω καλύτερα τι ρόλο μπορούν να παίξουν, με ποιο τρόπο μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο και πώς αυτές οι αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούσαν να αποτελέσουν συμμάχους για να μπορέσει να κλείσει θετικά αυτή η συμφωνία. Και το τρίτο τώρα. Τονίσατε ότι εδώ δεν πρόκειται βέβαια για ουσιαστικά εμπόδια όσον αφορά το κλείσιμο αυτών των συμφωνιών σχετικά με τόσα όσα αιτήματα έχει υποβάλει η Ινδία. Αν δεν είναι ουσιαστικά αυτά τα εμπόδια λοιπόν, πώς θα μπορούσε κανείς στη φάση αυτή, γιατί προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να βρούμε, να πετύχουμε το αποτέλεσμα που ευχόμαστε όλοι. Ποιο ρόλο ακριβώς θα έχει αυτό το πλησίασμα το πολιτικό, αυτή η προσέγγιση που παρατηρήθηκε σε αυτές τις προσπάθειες για ένα νέο διάλογο με την Κίνα. Ευχαριστώ. Η Μαρίτια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Πρέσβη. Τρεις σύντομες ερωτήσεις για το ΤΙΣΑ, την ε, Συμφωνία Συναλλαγών για, στον τομέα των υπηρεσιών. Συμμετέχουν πολλοί, έχουν μπλοκάρει οι Ηνωμένε Πολιτείε. Κάνει προσπάθειες ε, η Ένωση για να προχωρήσει η κατάσταση. Θα θέλατε το ΤΙΣΑ να μπει σε κάποιες πρωτοβουλίες του ΠΟΕ. Μπορεί να βοηθήσει ο ΠΟΕ να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Και τέλος, ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ προτάθηκε ως τρόπος για να αμφισβητήσουμε ε, αυτά που κάνει η Κίνα που μπλοκάρει το ίντερνετ και διάφορες άλλες οπτικοακουστικές. Η Κίνα έχει μπλοκάρει την πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες ε, αγορών των ΗΠΑ σε αυτόν τον τομέα. Θα μπορούσε μέσω του μηχανισμού επίλυσης διαφορών να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, γεια σας, ευχαριστώ. Για τον κύριο Πρέσβη, τις εξή ερωτήσεις για το 108 άρθρο του Συνθήκης Λισαβόνας. Τι λέει, ότι θα λάβει υπόψη αυτούς τους στόχους για την ανάπτυξη να εφαρμόσει τις πολιτικές που θα επηρεάσουν αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εμπορική σχέση θα πρέπει να λάβει υπόψη της και να έχει μια συνοχή, να δηλαδή, σχετικά με αυτή την ανάπτυξη να μειωθεί σύντομα η φτώχεια και αργότερα μακροπόθεσμα να την εξαφανίσουμε. Εδώ ε, δεν ξέρω, δεν εξυπηρετεί ε, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν τρομερές αντιφάσεις ανάμεσα στη συνεργασία για την ανάπτυξη και την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτο ερώτημα λοιπόν για τον κύριο Πρέσβη. Πώς, γίνεται ο συντονισμός από ε, τον με όσους εργάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη και αν συναντιέστε πόσο συχνά το κάνετε με τον επικοινωνία της ΕΦΚΟ. Λοιπόν, το δεύτερο ερώτημα τώρα. Πεστε μου κάτι σχετικά με, το, με την συμφωνία αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα Ηνωμένα Έθνη που θα εξυπηρετήσει να εξαφανίσει την ατιμορρησία για εγκλήματα από διάφορες εταιρείε και εδώ πέστε μας την άποψή σας τι κάνει σχετικά με τη μελλοντική συνθήκη τι κάνει την σχετικά με την αντιμορρυσία. Τι γίνεται με αυτές τις ε, υπηρεσίες που είναι, έχουν δραστηριοποιηθεί διεθνώς. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Πρέσβη για την παρουσίαση του. Το χειρότερο σκηνικό για αυτόν τον πολύπλευρο χαρακτήρα θα ήταν ο ΠΟΕ ακριβώς να παγώσει σχετικά με αυτή την ε, ε, συμφωνία. Είπε όμως και εδώ κανονικά υπάρχει μια πνοή κάποιες ε, ισοδοξίε ε, ότι υπάρχει ένα προσωρινό σχέδιο, πλαίσιο και θα ήθελα να μας πει τι είναι αυτό το το λογικό χρονικό πλαίσιο για να γίνει αυτό σχετικά με τον πολύπληρο χαρακτήρα. Και επίσης ε, ορισμένοι είπαν ότι τους ενδιαφέρει να υπάρχει ένα δεύτερο αναπληρωματικό σχέδιο ανάλογα με το υπάρχει αυτή η αναχέτηση στην ολυπορία του ΠΟΕ. Και ακριβώς ε, όσες ε, είπαν στην συμφωνία, ίσως τελικά να υπάρξει ε, μια κατάληξη που να μην συμπεριληφθούν δηλαδή όλα τα κράτη-μέλη, να μην συμμετάσχουν. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η πιθανότητα, νομίζω ότι είναι κάτι το λογικό. Και ακόμα κάτι. Η Κίνα προσπαθεί να πετύχει μια συμφωνία με την Ινδία. Η εκτίμησή σας είναι πώς θα μπορέσει να επηρεάσει μια παρόμοια συμφωνία σε αυτή την πολύπλευρη ε, συμφωνία, αυτή η συμφωνία μεταξύ Κίνας και Ινδίας. Ο κύριος Κατρούγκαλος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη, πώς αντιδράτε στις επικρίσεις για τον ΠΟΕ και για το ότι οι ερμηνείες που κάνει το σώμα προσφυγών γίνεται τελικά δημιουργούν ένα νομικό πλαίσιο που υπερισχύει της εθνικής νομοθεσίας ιδίως για τις ιδιωτικοποιήσεις και την απορρίθμιση. Ο Πρόεδρος, κύριε Πρέσβη, έχετε δυνατότητα τώρα να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, 8 λεπτά παρακαλώ. Ω, με συγχωρείτε. Κάποιον ξέχασα. Παρακαλώ. Παρακαλώ σύντομα. Και να δείχνετε την κάρτα σας, παρακαλώ, όταν ζητάτε το λόγο. Κύριε Πρέσβη. Οι διαπραγματευτές εργάζονται για το TTIP. Αν εγκριθεί θα είναι η μεγαλύτερη διμερή συμφωνία που έχει ποτέ υπογραφεί. Ακόμη και τώρα, χωρίς συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, οι εμπορικές σχέσεις είπα ενώσεις είναι περίπου ένα τρεις χρόνο. Θα είναι λοιπόν πολύ μεγάλη αυτή η εμπορική συμφωνία, πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε πρόσφατη. Εάν υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία, κατά τη γνώμη σας, τι επίπτωση θα έχει στο πολυμερέ σύστημα. Δηλαδή τι θα γίνει. Το Ντόχα έχει πεθάνει και το TTIP θα είναι απλώς ε, το φέρετρο. Πιστεύετε ότι το TTIP μαζί με το TPP είναι δείγμα ότι οι διμερείς συμφωνίες θα είναι οι πιο συνήθεις για το εμπόριο ή θεωρείτε ότι τόσο μεγάλες διμερείς συμφωνίες θα οθήσουν τις χώρες να συνεργαστούν πολυμερώς για να ελεγχθούν καλύτερα οι εμπορικές ροές εντός του ΠΟΕ. Έξι λεπτά κύριε Πρέδρε. Θίξατε πολύ σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Θα είμαι πολύ σύντομος, πρέπει να ακολουθήσω τις εντολές του Προέδρου. Ο Πρόεδρος ξεκίνησε λέγοντας ότι είμαι αισιόδοξο. Πολύ συχνά μου το λένε. Και η απάντησή μου είναι ότι όχι δεν είμαι αισιόδοξο. Εμείς ποτέ δεν πρόκειται να καταλήψουμε την πολυμερή προσέγγιση. Θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητε αξιοποίησή της. Γι' αυτό το λόγο στέλνω αυτό το μήνυμα και δεσμευόμεθα να ψάξουμε τέτοιες λύσεις. Υπό ιεσδήποτε συνθήκες. Η θητεία μου τελειώνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ελπίζω λοιπόν να κάνω απολογισμό αργότερα. Η Ένωση πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ένας πολύ θετικός παράγων, ιδιαίτερα αξιοσέβαστος, οι απόψεις μας γίνονται ακουστές και φυσιολογικά η λογική μας είναι λογική συμβιβασμών. Όχι, δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον κανόνα της ομοφωνίας. Κανείς δεν θέλει να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση. Απευθείας. Αλλά όλοι αναγνωρίζουμε ότι η πολυμερής προσέγγιση είναι πολύ ευέλικτη. Πολλές συμφωνίες που συνάπτει ο Πόεν είναι πολυμερείς χωρίς να θέτουν ένα αμφιβόλο την ομοφωνία. Το θέμα είναι λοιπόν να εφαρμόζεται όλο και περισσότερο η πολυμερής προσέγγιση. Και αυτή η πορεία προς ε, την πολυμερή προσέγγιση ήδη συμβαίνει, όπως μέσω της ΤΙΖΑ, του ITA, των συμφωνιών για τα περιβαλλοντικά αγαθά. Κερδίζει λοιπόν όλο και περισσότερο η πολυμερής προσέγγιση. Έχει προχωρήσει πολύ η εργασία για την ΤΙΖΑ, τη Συμφωνία για Συναλλαγές ε, στον τομέα των υπηρεσιών. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι η Κίνα. Και ο Ζαν Λουκ είπε σήμερα το πρωί ότι είμαστε και το έχουμε πει ανοιχτά υπέρ της ε, ένταξης της Κίνας. Αλλά η Κίνα Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες άλλων για τις συνθήκες συμμετοχής της στις διάφορες πολυμερείς διαπραγματεύσεις. Και τώρα είμαστε σε φάση, κρίσιμη φάση διαπραγματεύσεων για την επέκταση του ITA, και θετικά έχει συμμετάσχει η Κίνα στις προσπάθειες για τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά. Θέλω να είμαι πολύ καθησυχαστικός για αυτούς που είπαν ότι η Ένωση δεν ενδιαφέρεται πια για την πολυμερή προσέγγιση. Μα το είπα και στην παρουσίασή μου. Η πολυμερής προσέγγιση είναι η κύρια προτεραιότητά μας. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου συλλογικά, πολυμερός, δεν επιτυγχάναμε αποτελέσματα καιρό τώρα. Όπως είπα, κάθε φορά που κάτι μπορεί να επιτευχθεί πολυμερός, προσπαθούμε να το επιτύχουμε. Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε το προσωπικό, έχουμε τους πόρους να πιέσουμε για πολυμερείς λύσεις όπου ρεαλιστικά είναι εφικτές. Ο Παύλο είπε μια πολύ σωστή ερώτηση. Θα απαντήσω σύντομα. Έχουμε την Ινδία και αυτή την σύνδεση μεταξύ της δημόσιας ε, αποθήκευσης και της διευκόλυνσης του εμπορίου. Αυτή η δυσχέρεια μπορεί να είναι καταστροφική, αλλά αν την υπερβούμε και περάσουμε σε πολυμερή προσέγγιση, θα έχουμε μεγάλες προκλήσεις για να καταλήξει το DTA. Αυτό, πιστεύω, θα είναι η κύρια πρόκληση. Η αντιμετώπιση των αναπτυσσόμενων χωρών. Πολλά υπόθηκαν γι' αυτό. Ο ΠΟΕ, πρέπει να πω, είναι ο πιο δημοκρατικός διεθνής οργανισμός που υπάρχει. Δεν υπάρχει διευθυντήριο, δεν υπάρχει συμβούλιο ασφαλεία, ο καθένας έχει μία ψήφο, ο καθένας έχει ίσο χρόνο ομιλίας, ο καθένας έχει τον ίδιο χώρο για να λειτουργήσει, πολύ μικρό ε, και πολλές χώρες ε, μπορεί να είναι μικρές αλλά επειδή δουλεύουν αποφασιστικά κάνουν πολύ έργο στον ΠΟΕ η Ένωση επίσης εργάζεται θετικά στα πλαίσια του που Έχουμε βοηθήσει να λυθούν πολλά θεμελιώδη θέματα και στις διαπραγματεύσεις του Μπαλί για τους κανόνες προέλευσης. Ό,τι είναι σε αυτές αποφάσεις οφείλονται και στη συμβολή της Ένωσης ε, που συνέβαλε θετικά και αντιμετωπίζεται και ως θετικά συμβάλλουσα. Η Ινδία θα μπορούσε να βοηθήσει και ελπίζω να το κάνει. Αυτό που είπα για την ουσία, το είπατε δύο-τρεις φορές, τα αιτήματα της Ινδίας ε, αφορούν και την ουσία για αυτή την ε, δημόσια αποθήκευση και επιστηστική ασφάλεια που έχει ανησυχίες για αυτά τα θέματα η κυβέρνηση της Ινδίας και είναι πολύ ουσιώδες συζητήσεις. Αυτό που είπα είναι ότι το συνδέουν με την διευκόλυνση του εμπορίου και αυτό είναι θέμα τακτικής. Είναι πολιτική επιλογή. Και γι' αυτό είπα ότι για να υπάρξει πρόοδος πρέπει να είμαστε βεβαίως ευέλικτοι αλλά να σεβαστούμε τα πορίσματα του Μπαλί. Δηλαδή η διευκόλυνση εμπορίου πρέπει να προχωρήσει. Και το χρονοδιάγραμμα είναι, είπα, θέμα εβδομάδων. Έχουμε συναντήσεις του ΠΟΕ που κάθε μέρα κάνουν το κλίμα πιο τεταμένο είναι σαφές ότι δεν μπορεί να ε, προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις εάν δεν υπάρξει ένα ξεμπλοκάρισμα της κατάστασης. Γιατί αλλιώς ε, θα αυξηθούν οι εντάσεις, ε, θα φτάσουμε σε περιβάλλον κρίσης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση. Εάν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση, πιστεύω ότι θα βελτιωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οι αναπτυσσόμενες χώρες πολλά υπόθηκαν για αυτές, αλλά νομίζω ότι έχω απαντήσει συνολικά, δεν θα επαναλάβω. Τίζα, όπως είπε και ο Ζανλουίκ Είμαστε υπέρ της συμμετοχής ε, της Κίνας στην Τίζα, αλλά συνδέεται και με τα άλλα βήματα για διάφορα πολυμερή θέματα που πρέπει να υπάρξουν τους επόμενους μήνες. Έχουμε ένα σχέδιο, σχέδιο Β, για να αποφύγουμε το πάγωμα. Ανάφερα κάτι, δεν είναι όμως εναλλακτικό σχέδιο, είναι η δυναμική της κατάστασης ή θα καταφέρουμε να ξεπαγώσει η κατάσταση, να υπάρξει κινητικότητα, να επανέλθουμε στην πολυμερή μέθοδο ή ο θα ξεκινήσει μια συζήτηση για μια πολυμερή επιλογή για την ε, διευκόλυνση του εμπορίου και μια ευρύτερη συζήτηση για το τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό για τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστεί ο οργανισμός στο μέλλον γιατί θα είναι μια πολυμερής λύση για αυτό που είναι η ουσία της συνολικής προσέγγισης του ΠΟΕ. Γιατί αυτό είναι και το πόρισμα του Μπαλί. Εάν αυτό το πόρισμα μετατραπεί σε μια συζήτηση για πολυμερείς λύσεις, θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις για την οργάνωση. Και τέλος, τέλος, ένα λεπτάκι ακόμη. Το θέμα του TTIP. Υπόθηκαν πολλά για το εάν θα προτιμηθεί η, πολυμερής, η δίμερη συγγνώμη, προσέγγιση. Κοιτάξτε. Θα πω αυτό που είπε και ο Ρομπέρτο ε, Αθεβέδο, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ, με τον οποίο έχω, έχω συνεργαστεί αρκετά χρόνια, που σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο για πολλά θέματα. Ή είπε ο Αθεβέδο ότι πρέπει να έχουμε την εικόνα μιας πυραμίδας. Τα θεμέλια και το πρώτο επίπεδο είναι η πολυμερής προσέγγιση και το διμερές χτίζει πάνω σε αυτό. Βεβαίως διμερός ε, κάποια συμβαλόμενα μέρη μπορούν να φτιάξουν περισσότερους κανόνες συμβατότητας ε, φιλελευθεροποίησης. Αλλά βασιζόμενοι στο παρακάτω. Να έχουμε λοιπόν αυτή την εικόνα ότι οι προκλήσεις της ε, εμπορική πολιτικής είναι σαν πυραμίδα. Βάση πολυμερει κανόνε κανόνες επί των οποίων εδράζονται περαιτέρω οι ε, διμερείς προσπάθειες που αυξάνουν την συμβατότητα, αυξάνουν ε, την προσπάθεια αναρμόνισης ε, των προδιαγραφών και κανόνων. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να είναι ο στόχος μας. Αυτή είναι η μόνιμη πρόκληση έτσι πρέπει να το δούμε. Συμβάλλουν και τα δύο. Και οι πολυμερείς προσπάθειες και οι διμερείς, αλλά όλα αυτά πρέπει να συμβάλλουν στην επόμενη φάση πολυμερών διαπραγματεύσεων. Με συγχωρείτε, ίσως δεν απάντησα σε όλα, αλλά νομίζω ότι απάντησα σε αυτές που ε, ήταν ε, μέλημα ε, περισσότερων βουλευτών. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Δεν είναι πιστεύω τελευταία φορά που θα είστε ενώπιόν μας και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Και τώρα τελειώσαμε με αυτό το θέμα της μέλισσας διάταξης και περνάμε στο 11 το οποίο είναι η ψηφοφορία. Ελπίζω λοιπόν να έχετε όλοι τις ε, κάρτες σας γιατί οι ψηφοφορίες θα γίνουν ηλεκτρονικώς. Ψηφίζουμε το πρωτόκολλο για την Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Κορέας λόγω της ένταξης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συγητής είναι ο κύριος Ζάντι. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε αυτή τη σύσταση. Παρακαλώ ψηφίστε. Πρώτα απ' όλα να ελέγξουμε εάν είναι όλοι παρόντες και αν αντιστοιχούν στον αριθμό μελών που αντιστοιχεί στην πολιτική τους ομάδα και μετά θα ε, γνωστοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Για τη σύσταση του κυρίου Σαχράντιλ. Πέρα της ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα. ...33 υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον Σύντη. Οπότε, σύντομη ήταν η πληροφορία σήμερα. Τελειώσαμε και με το 11. Και περάμε στο 12. Το θέμα των επιπτώσεων των κυρώσεων που εφαρμόζονται στα πλαίσια της ε, σύγκρουσης Ένωσης Ρωσίας. Επανειλημμένα έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Τι οικονομικές επιπτώσεις έχουν αυτές οι κυρώσεις. Και θα πρέπει και πάλι να επιχειρήσουμε να έχουμε και επιστημονικές συμβουλές γι' αυτό. Χαίρομαι λοιπόν που είναι παρόν ο κύριος Μάικλ Έμεσον για το Κέντρο Ευρωπαϊκών ε, Σπουδών. Χαίρομαι που είναι μαζί μας. Τον καλωσορίζω για να ε, θέσει τις βάσεις για τη συζήτησή μας. Και του δίνω το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου τιμή που με καλέσατε ε, να συμμετάσχω στη συζήτηση αυτή. Ε, ε, μέσω της γραμματείας έχω διανύμει στα, έγγραφα, στα μέλη ένα έγγραφο το οποίο αφορά κάποια στοιχεία τα οποία θα αναφέρω εδώ. Πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Υπάρχουν νέα βάση ενός, μιας νέας επιστολής από τον Πούτι στον Ποροσέγκο που ρίχνει λίγο φως ε, στις αντιδράσεις ε, της ε, Ρωσίας, αλλά θα επανέλθω αργότερα θα διαρθρωθεί ως εξής η παρέμβασή μου. Κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τις κυρώσεις από τη μία πλευρά μετά τις κυρώσεις από την άλλη καθώς επίσης και το θέμα της υλοποίησης της Συμφωνίας Σύνδεσης και πως ε, ε, οι κυρώσεις ε, ε, σχετίζονται με τη συμφωνία αυτή. Οι κυρώσεις συνήθως ε, δεν έχουν ε, καθόλου καλό αποτέλεσμα. Έχουμε παρόμοιες περιπτώσεις σε διάφορες υποθέσεις, αλλά βεβαίως υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή του Σμπεκιστάν που οδήγησαν σε κάποιες θετικές ας πούμε εξελίξεις. Υπάρχουν και οι κυρώσεις οι οποίες έχουν μετριασμένα αποτελέσματα. Αυτά έχουν μελετηθεί ως, έχοντες, ως έχουσες αποτέλεσμα της τάξης του 5%. Άκουσα προηγουμένως με πολύ μεγάλο ε, ενδιαφέρον και τον ε, ε, αντιπρόσωπο των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένα Έθνη που θεωρεί ότι η κυρώσεις είναι πάρα πολύ δημοφιλής και θα συμφωνήσω στην απάντηση που δίνει γιατί όταν κανείς αντιμετωπίζει αντιμετωπίζει έναν προβληματικό ε, εταίρο ε, δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα από τα λόγια και τον ε, πόλεμο. Εδώ ισχύει ιδιαίτερα στην Ουκρανία γιατί βεβαίως η Ρωσία προχώρησε σε πολεμική σύγκρουση. Εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο φυσικά. Τώρα, Πού οδηγούμαστε. Οδηγούμαστε συχνά στο ότι οι κυρώσεις αποτελούν πολιτική δήλωση σημαντικές πολιτικές ε, δηλώσεις οι οποίες όμως είναι αποσυνδεδεμένες από, ε, από τον ουσιαστικό αντίκτυπο ε, που μπορεί να έχουν κάποιες σοβαρές πολιτικές δηλώσεις οι οποίες διασφαλίζουν κάποια ελάχιστη διασύνδεση ανάμεσα στα λόγια και τις στην εσωτερική συζήτηση. Αυτές ήταν λοιπόν οι κατηγορίες προηγουμένως. Είπαμε ευρωπαϊκές ενωσιακές κυρώσεις κατά της ε, Ρωσίας οι οποίες αφορούν ε, οικονομικές κυρώσεις καθώς επίσης και διπλωματικές που αφορούν δηλαδή ε, το διπλωματικό προσωπικό. Είναι αυτές οι οποίες συζητήθηκαν σε επίπεδο διασκέψεων κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι εγώ παρακολουθώ από πολύ στενά και τα όσα αναφέρουν στον ρωσικό τύπο και επομένως από πολιτική άποψη δεν ε, ε, ενοχλείται και πάρα πολύ ο Πούτιν από αυτές τις ε, κυρώσεις από πλευράς των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης δεν είδαμε και από πλευράς των G20 να υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να επιβεβαιωθούν ας πούμε, να επιβεβαιωθεί το βάρος των κυρώσεων. Ξέρουμε επίσης πως έχει η κατάσταση στην Κρυμαία και μετά στο Λουγκάν και στο Ντονιέσκ. Πρέπει να το δούμε καθαρά το θέμα αυτοί που υφίστανται τις κυρώσεις ε, και ε, οι Ρώσοι θεωρούν ότι αυτά είναι παράσημα, αυτές οι κυρώσεις είναι ε, παράσημα στο στήθος τους και επομένως πραγματικά έχει αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο. Οι οικονομικές κυρώσεις τώρα, αυτές είναι λίγο πιο σημαντικές, πάυση δραστηριοτήτων όσον αφορά την τράπεζα ανασυγκρότηση, όσον αφορά το EB, αυτό είναι πιο σημαντικό σημαντικό και ε, ε, ε, έχει αντίκτυπο και στην πρόσβαση που έχουν οι ρωσικές τράπεζες στην διεθνή, στην παγκόσμια αγορά. Βεβαίως η Ροσνεφτ, η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία, πρέπει να βρει 15 εκατομμύρια έτσι ώστε... Ε, πρέπει να βρει 40 δις έτσι ώστε να μπορέσει να ξεπληρώσει ε, τις υποχρεώσεις απέναντι στις διεθνείς ε, τράπεζες. Αυτό είναι βέβαια πολύ ενδιαφέρον και για μας γιατί προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στο establishment το, οποίο, το, τραπεζικό το Κρεμλίνο και οι άλλες ε, ε, ε, υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν την κατάσταση απλώς έβγαλαν τον Τουσέγκο από την από, από τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει από την πλευρά ε, των ε, Γάλλων υπάρχει και μία άλλη υπόθεση των Μιστράλ ε, και αυτό είναι ένα πολύ θεαματικό γεωπολιτικό πρόβλημα. Είναι αυτό γκολ το οποίο έχει ρίξει αυτή τη στιγμή η Γαλλία όσον αφορά την, την υπόθεση των πλοίων Μιστράλ. Όσον αφορά τώρα τα αντι, τις αντικυρώσεις νομίζω ότι κάποιος από τη Γενική Διεύθυνση έκθεση Γεωργίας ε, αναφέρθηκε σε αυτό. Πάντως οι υπολογισμοί μου είναι ε, ότι οι εξαγωγές είναι ένα περίπου της 100 του ΑΕΠ, ενώ ε, τη πλευρά της Ρωσίας είναι ένα δέκατο του ΑΕΠ. Ε, είναι επομένως από ε, μακροοικονομική άποψη, είναι πολύ μικρό το στοιχείο, έστω και αν είναι ιδιαίτερα προβληματικό για ορισμένους. Βεβαίως από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρουμε ότι μακροοικονομικά το κλίμα, το μακροοικονομικό κλίμα θα υποστεί ε, μια αρνητική ε, τροπή. Παρόλα αυτά ε, δεν φαίνεται να δημιουργούνται ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα για την ώρα και εν πάση περιπτώσει αυτό εντάσσεται στο πρόβλημα του τρόπου με τον οποίο θα αντιμετωπίσει το θέμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην συνεργατική της πολιτική. Τρίτο, ίσως φαίνεται ελάσσονο σημασία, αλλά κατά την άποψή μου είναι το πιο σημαντικό. Ε, δηλαδή είναι ε, το γεγονός ότι ήδη η Ρωσία ε, τιμωρεί την Ουκρανία και τη Μολδαβία, όπως έκανε στο παρελθόν και με τη Γεωργία, με πάρα πολλές ε, κυρώσεις. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και προχωράει με φυτοϊγειονομικούς περιορισμούς, που βεβαίως έχουν καθαρά πολιτική χρειά threatens. Και τώρα η Ρωσία επιπροσθέτως απο, απειλεί την ε, ε, Ουκρανία ε, να διαγράψει το πρωτομισιακό καθεστώς για μια σειρά προϊόντων. Έγινε την προηγούμενη πέμπτη μια ε, συνεδρίαση, μια συνάντηση κατά την οποία ο Επίτροπος Ντεχούχτ εξ ονόματος Επιτροπής ε, συμφώνησε ε, να μεταθέσει την το, το, το προτιμησιακό εμπορικό κομμάτι της γενικότερης συμφωνίας και βεβαίως αυτή δεν είναι μια απόφαση που μπορεί να πάρει μόνος του θα πρέπει να την υποβάλει στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα πάρει θέση από αυτού έτσι οδηγούμαστε σε αυτήν την μεταβατική περίοδο, πριν δηλαδή αποφασίσει τη θέση του το Συμβούλιο, σε μια σειρά καταστάσεων. Αμέσω μετά την συνεδρία αυτή, ο Λουκάγεφ, ο Υπουργό έστειλε, Ρώσος Υπουργός έστειλε μια επιστολή στον ε, Επίτροπο Ντεγκούχτο, ε, και μάθαμε σήμερα το πρωί ότι έστειλε και μια άλλη επιστολή στο, τον Ποροσέγκο την οποία διαβάσαμε στον τύπο, διέρευσε δηλαδή στον τύπο. Εκεί λοιπόν λέει ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, για αυτήν την ε, παραχώρηση αλλά εμείς θέλουμε πολλά περισσότερα. Ε, Ιδίω δε η Ρωσία αναφέρει ότι, μάλλον ο Πούτιν λέει, ότι εάν η Ουκρανία αρχίσει να προετοιμάζει την εφαρμογή του DCFTA, ε, Deep Comprehensive Trade Agreement, ε, τότε ε, εμείς μπορεί να πάρουμε κάποια άλλα αντίμετρα. επομένω αυτό το οποίο αρχικά καλή την πίστη δέχτηκε ο Επίτροπος Gucht, δηλαδή μια, μια χείρα βοηθείας ας πούμε διαπραγμάτευσης έτσι ώστε να λυθούν κάποια προβλήματα, προφανώς Ρωσία το εκλαμβάνει ε, διαφορετικά. Εν συμπεράσματι κύριε Πρόεδρε ε, μπορώ να πω ότι οι οικονομικές κυρώσεις ε, κατά της Ρωσίας είναι σημαντικές αλλά δεν αλλάζουν ε, ε, την πολιτική υπό το φως της ε, τεράστιας προσπάθειας της προπαγάνδας που κάνει η ρωσική πλευρά που έχει οδηγήσει τελικά το, την ρωσική κοινή γνώμη σε πολύ γενικές γραμμές να λέει ότι εμείς θα υποφέρουμε αρκεί να μην περάσουν οι φασίστες που τους στηρίζουν, που τους στηρίζουν οι Ευρωπαίοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η αφήγηση την οποία έχουν περάσει στους περισσότερους ε, ε, ε, Ρώσους. Αυτή είναι η αφήγηση που κατανοούν οι Ρώσοι που βεβαίως είναι αφρικτό ψέμα αλλά παρόλα αυτά έτσι είναι. Επομένως σημαντικές συγκυρώσεις αλλά δεν έχουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Επίσης τα ρωσικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται κατά της Ουκρανίας και ενδεχομένως κατά και της Μολδοβίας γιατί μιλάμε τώρα για τις για την Ουκρανία, αλλά τα τέλη Νοεμβρίου έχουμε και τις εκλογές στην ε, Μολδαβία και επομένως ε, θα δούμε τι θα γίνει εκεί όσον αφορά ε, τους φιλορώσους πολιτικούς. Αυτές λοιπόν ε, οι τελευταίες ε, πρόσφατες ε, εξελίξεις αποτελούν σημαντική απειλή για το γενικότερο οικοδόμημα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και για την εξέλιξη. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στο μόνιμο εισηγητή μας για τη Ρωσία. κύριος Βέιν. Ο κύριος Ρέν, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Έμεσον για την πολύ σωστά τοποθετημένη και πολύ ρεαλιστική εκτίμησή του των επιπτώσεων των κυρώσεων. Να θέσω δύο-τρεις περαιτέρω ερωτήσεις στον κύριο Έμεσον για τις κυρώσεις αυτές και τις επιπτώσεις τους. Όπως είπατε, οι κυρώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι οι πιο ουσιώδεις. Αυτό το είπε και ο Αλεξέη Κούντριν, ο πρώην ε, Υπουργός Οικονομίας, που ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους ε, Υπουργούς Οικονομίας στον κόσμο την παρελθούσα δεκαετία. Σε αυτό το πλαίσιο ερωτώ πώς θεωρείτε ότι θα επιδράσουν αυτές οι κυρώσεις στις ρωσικές τράπεζες στο εγγύς μέλλον τις δυνατότητές τους δηλαδή αναχρηματοδότησης μεγάλων εταιριών στη Ρωσία. Και τι επιπτώσεις θα έχει στον κλάδο του πετρελαίου και τις αναγκαίες επενδύσεις που χρειάζονται για τεχνολογική εξέλιξη του τομέα. Τι επιπτώσεις θα έχει εάν οι κυρώσεις παραμείνουν πάνω κάτω όσο έχουν αυτή τη στιγμή. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα της ε, ευρωπαϊκής εξάρτησης ενεργειακής εξάρτηση και θα έπρεπε να είναι το αποφασιστικό βήμα για να αυξήσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια. Βέβαια, ενώ εμεί μιλάμε για ανεξαρτησία από την Ανατολή, στη Ρωσία συζητούν ανεξαρτησία από τη Δύση. Οπότε, πώ βλέπετε αυτή την κατάσταση, μια που ξέρετε τόσο καλά τι συζητιέται στη Ρωσία, τι πολιτική μπορούμε να αναμένουμε και για το πετρέλαιο και για το φυσικό αέριο. Γιατί σε μεγάλο βαθμό δεν έχει αναφερθεί ως όπλο των ε, αντικυρώσεων. Τρίτη ερώτηση. Ίσως κάνουμε χωριστή συζήτηση για τα γεωργικά θέματα και το συζητήσαμε ήδη στην Επιτροπή Γεωργίας. Αλλά Στον τομέα αυτό χρειάζεται αλληλεγγύη μεταξύ ημών για να αντιμετωπιστούν οι ρωσικές αντικυρώσεις, τα αντίμετρα, γιατί έχουν επιπτώσεις τα αντίμετρα σε συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνίας. Και είναι ουσιώδες αν συνεχίσουμε αυτές τις κυρώσεις ε, να εξακολουθήσουμε να έχουμε την ε, στήριξη του πληθυσμού μας. Αυτά τα ερωτήματα στον κύριο Έμερσον. Και τώρα οι πολιτικές ομάδες για το ΕΛΚ. Ο κύριος Βάλης. Ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Διάβασα όλα τα στοιχεία για αυτή την ε, παρουσίαση. Είπατε ότι δεν είναι αποτελεσματικές οι κυρώσεις. Το να πει κανεί πώ ε, λειτουργούν οι κυρώσει, το να πει κανεί ότι δεν έχουν αποτέλεσμα οι κυρώσει, δείχνει πως δεν καταλαβαίνουμε πως λειτουργούν. Γιατί η αποτελεσματικότητά τους πρέπει να μετράτε σε σχέση με το ποιος θεωρούμε ότι είναι ο στόχος τους. Το να μιλάμε για αποτελεσματικότητα των κυρώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο και μετρήσιμο στόχο που υποτίθεται πως έχουν οι κυρώσεις. Και οι κυρώσεις δεν έχουν ένα σαφή μετρήσιμο στόχο. Ρωσία για παράδειγμα. Ποιος είναι ο στόχος των κυρώσεών μας προς τη Ρωσία να επιστραφεί η Κρυμαία στην Ουκρανία ή να αποφευθεί η πλήρης ε, προσχώρησή της στη Ρωσία ή να παραμείνει ε, ως υπανάπτυκτη περιοχή της Ρωσίας που θα δημιουργήσει προβλήματα ή να παρεμποδίσουμε τους Ρώσους από το να καταστρέψουν ε, εντελώς την Ουκρανία ή να αποτρέψουμε την προσάρτηση μεγάλων περιοχών της Ανατολικής ή και όλης της Νότιας Ουκρανίας ή να σταματήσουμε τη ρωσική στήριξη για τις αποσχιστικές ε, δυνάμεις στο Λουγκάνσκ και στο Ντονιέτσκ. Να πεντέξει διαφορετική διαφορετικοί Και ανάλογα με τον καθένα θα έπρεπε να μετρηθεί και η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων. Τι εννοώ. Οι κυρώσεις δεν έχουν ένα στόχο. Ο μόνος του στόχος είναι πρώτον να πληρώσει κάτι ο εισβολέας και ήδη πληρώνουν οι Ρώσοι παρά το πόσο περιορισμένες είναι οι κυρώσεις. Και δεύτερον, δεύτερος στόχος είναι να το ξανασκεφτεί ο εισβολέα πριν υπάρξει, πριν επιχειρήσει κλιμάκωση. Και η κατάπαυση του πυρός είναι μία απόδειξη ότι το λαμβάνουν υπόψη οι Ρώσοι, επιπλέον οι κυρωσει Είναι ένα μόνο από τα όπλα στη φαρέτρα της εξωτερικής πολιτικής. Ένα μόνο από τα βέλη. Από μόνο του δεν μπορεί να ε, οδηγήσει σε επιτυχία ή να θεωρηθεί υπεύθυνο για την αποτυχία. Και πρέπει να πω ακόμη ότι εκπλήσωμε. Διότι έχουμε ήδη παραδείγματα κυρώσεων. Και πώς υποτίθεται πως δεν λειτουργούν. Παραδείγματα. Μιανμάρ, Βυρμανία. Τα τελευταία χρόνια η χώρα αυτή έχει σημειώσει μεγάλες πρόοδους. Τόσο πολύ που οι κυρώσει μα ήρθησαν το 2013. Είναι τρομερή επιτυχία. Δεύτερον, Ιράν. Για πρώτη φορά, εδώ και πολύ καιρό, οι Ιρανοί προσήλθαν ε, στη Βιέννη και διαπραγματεύονται τις πυρηνικές τους βλέψεις. Ποτέ δεν θα είχε διαπραγματευτεί το Ιράν αν δεν είχαν επιβληθεί κυρώσεις γιατί υπήρξαν πολύ βαριές κυρώσεις στο Ιράν και μείωσαν τη δυνατότητά του να αποκτήσει τα αναγκαία υλικά για το πυρηνικό πρόγραμμα και γονάτισαν την οικονομία του. Αν δεν είχαν υπάρξει κυρώσεις θα είχαν προχωρήσει πολύ περισσότερο το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Ορίστε, επιτυχίες. Αλλά υπάρχουν και άλλες επιτυχίες. Η κατάργηση του Apartheid ε, στην Νότια Αφρική, η περίπτωση της ακτής ελεφαντοστού λοιπόν. Καλό όλε τι πλευρέ να είναι πιο προσεκτικέ όταν συζητάνε την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων. Να μην επιτρέψουμε ε, σκέψει που δεν ε, είναι σωστέ να μα παρεμποδίζουν από το να καταλήγουμε σωστά συμπεράσματα. Βίκτορ. Ευχαριστώ. Πολύ καλό να ακούμε τη γνώμη ειδημόνων, επιστημόνων. Μπορούν να βοηθήσουν τους πολιτικούς να καταλήξουν σε σωστά συμπεράσματα. Να δουν σε βάθος τα προβλήματα που είναι το πρόβλημα, οι στρατηγικές μας, οι σχέσεις με τη Ρωσία. Βεβαίως δεν θέλουμε να κάνουμε πόλεμο. Δεν θα ήταν λύση να κάνουμε πόλεμο εμείς με τη Ρωσία. Αλλά οι κυρώσεις είναι από πολιτική άποψη πολύ σημαντικές για την Ένωση. Να μην αποδεχθούμε τα τετελεσμένα που επιβάλλουν τρίτη είτε η Ρώσια είτε άλλοι. Ποτέ δεν πρέπει να παραδιδόμεθα αμαχητή, να αποδεχόμεθα τετελεσμένα όταν έχει κατάφορα παραβιαστεί ο διεθνής νόμος όπως την Κρυμαία και κατόπιν μέσω αυτού του πολέμου κατά της Ουκρανίας. Δεύτερον, υπάρχει οικονομική διάσταση. Αναφέρθηκε σαφώς για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, για τις δυσχέρειες που έχουν οι μεγάλες ρωσικές επιχειρήσεις ή η αποσύνδεση της, ε, διπλής, των τεχνολογιών διπλής χρήσης. Είναι απαράδεκτο για τις αξίες μας ως ευρωατλαντική οικογένεια να διαπιστώνουμε ότι ένας εισβολέας ωφελείται με τον ίδιο τρόπο από, διάφορα, από διάφορες δυνατότητες όπως εμείς. Και επίση τι άλλη εναλλακτική λύση έχουμε εκτός από κυρώσει. Δεν έχουμε άλλες. Μόνο κυρώσει. Αν είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε, να την αξιοποιήσουμε. Σοβαρά, αποτελεσματικά, συνεπέστερα. Χαίρομαι που αναφέρθηκε το θέμα των ε, φρεγατών Μιστράλ. Βεβαίω, εμεί οι Ευρώποι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν είναι θέμα ότι μόνο η κεντρική και ανατολική Ευρώπη έχει να φοβηθεί από τη Ρωσία. Είναι μια πρόκληση για όλους μας. Και πρέπει λοιπόν να είμαστε όλοι συνεπεί και ενωμένοι. Και για να βελτιωθεί η στάση μας είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η ευρωατλαντική σχέση. Να αναφερθούμε βεβαίως στα αποτελέσματα της συνάντησης στο Newport. Βεβαίως υπάρχουν διάφοροι που παπαγαλίζουν την ρωσική προπαγάνδα αλλά δεν θέλουν να ακούσουν αυτά που λέω τώρα. Επιπλέον η Ευρώπη πρέπει να αρχίσει να αυξήσει, να αρχίσει να οικοδομεί τις αμυντικές της δυνατότητες. Ο πρόεδρος Ολάντ ε, είπε ότι δεν πρέπει να εξαρτώμεθα πλήρως από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να αναπτύξουμε τις δικές μας δυνατότητες. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε. Να το επιτύχουμε αυτό. Και τέλος, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε ουσιώδη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης για θέματα ασφάλειας και άμυνας. Διότι αυτή τη στιγμή οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης εξαρτώνται από τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ και αυτό είναι επιζήμιο για την ενωσιακή αλληλεγγύη. Ως Ρουμάνος βεβαίως τονίζω ότι πρέπει να μας βοηθούν οι στρατιωτικές δυνατότητες ε, της Ένωσης και όχι μόνο του ΝΑΤΟ, χωρίς βεβαίως να αντιτίθενται αυτές οι δύο μεταξύ τους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπείς και να συνεχίσουμε να πιστεύουμε και τι ευρω ατλαντικές μας αξίες. Για το ECR, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα επανέλθω στα εμπορικά θέματα που νομίζω πως είναι το κύριο θέμα για μας. Δύο σύντομες ερωτήσεις για τα ρωσικά αντίμετρα κατά της Ένωσης. Να διευκρινίσω μερικά στοιχεία. Πρώτον, αυτά τα αντίμετρα αφορούν μόνο εξαγωγές τροφίμων. Κρέας, προϊόντα κρέατος, ε, γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά, ψάρια και άλλα. Υπάρχουν τίποτε άλλα προϊόντα που επηρεάζονται από αυτά τα αντίμετρα. Και δεύτερον, τώρα για τα συγκεκριμένα στοιχεία. Βλέπω εδώ στο κείμενο του κυρίου Έμερσον ότι οι εξαγωγές ε, αγροτροφημικών είναι 12 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι 0,09 του ΑΕΠ της Ένωσης. Ενώ στο δικό μας έγγραφο λέγεται, εδώ ΝΑΤΟ, είναι ότι τα προϊόντα τα οποία αφορούν τα αντίμετρα είναι μόνο 43% των ε, γεωργικών μας εξαγωγών προς τη Ρωσία, το οποίο είναι 5,1 δις, όχι 12. Και το ποσοστό του ενωσιακού ΑΕΠ είναι κάτω από το μισό από αυτό που λέει το κείμενο του κυρίου Έμερσον. Το αποτέλεσμα των κυρώσεων λοιπόν, αν δεν καταλαβαίνω καλά, είναι 0,045 του ενωσιακού ΑΕΠ. Είναι σωστό αυτό. Αυτό λέει το δεύτερο κείμενο. Και κάτι τελευταίο. Στο σημείο 6 αυτή η έκθεση για την τριμερή συνάντηση Κομισιόν Ρωσία-Ουκρανία την οποία επέκριναν κάποιοι συνάδελφοι. Όχι, δεν νομίζω ότι πρέπει να επικρίνουμε αυτή τη συνάντηση. Νομίζω ότι ήταν ένα δείγμα της καλής διάθεσης της πλευράς μας ότι είχαμε κάθε καλή διάθεση να βρούμε κάποια αποδεκτή λύση χωρίς να θυγεί ούτε η Ουκρανία ούτε η Ένωση. Οπότε δεν θέλω να επικρίνω αυτή την προσέγγιση πρέπει να την ε, εκτιμήσουμε ρεαλιστικό, με ρεαλιστικό τρόπο. Ο Χέλμουτ. Ευχαριστώ Μπέρντ. Είμαστε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο της συζήτησης. Είμαστε Επιτροπή Εμπορίου εδώ, που ασχολείται με την οικονομική πλευρά της πολιτικής κυρώσεων από κάθε άποψη επιπτώσεις των κυρώσεων για την Ένωση και για την ε, Ρωσία των εκατέρωθων κυρώσεων στα πλαίσια της γενικότερης βεβαίως πολιτικής μας στρατηγικής. Κατά τη γνώμη μου, δεν το είπαμε σαφώς στους ειδικούς. Ο εμπειρογνώμων λέει ότι μόνο στον τομέα της γεωργίας αφορά ε, ένα έως τρεις τομείς συγκεκριμένους. Αλλά αυτό αφορά και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και σε εμά και στη Ρωσική Ομοσπονδία. Δηλαδή, εάν ορισμένες... Ε, εάν ορισμένα προϊόντα κρέατος ή γαλακτοκομικά προϊόντα δεν πολλούνται εκεί που επολούνται, αυτό έχει ως επίπτωση ανεργία, ή και κατάρρευση, πτώχευση των επιχειρήσεων που θα έκαναν αυτές τις ε, εμπορικές συναλλαγές. Γιατί τέθηκε το ερώτημα, ποιος είναι ο στόχος των κυρώσεων. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Στόχος των κυρώσεων της Ένωσης είναι να συμβάλλει μεσοπρόθεσμα και, βράχη πρόθεσμα να επιδεινωθεί η κατάσταση της κοινωνίας ε, στην Ρωσική Ομοσπονδία. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρξουν αλλαγές και στην ε, πολιτική κατάσταση. Ή είναι στόχος των κυρώσεων να έχουν ένα άμεσο ταχύ αποτέλεσμα για να αλλάξει η πολιτική της Ρωσίας έναντι της Ένωσης. Και τώρα νομίζω ότι είμαστε δέσμοι της δικής μας λογικής. Γιατί δεν έχουμε καμία λογική. ξεκινάμε αυτές ε, τις κυρώσεις χωρίς να έχουμε μέσο και μακροπρόθεσμη προοπτική. Στη Γερμανία οι οικονομικοί κύκλοι ε, έχουν μεγάλες ανησυχίες για τις ε, προοπτικές αυτές. Για παράδειγμα, μια εταιρεία στο Βερολίνο, η MRN, ήδη ανήγγειλε μειωμένα ωράρια εργασίας για διάφορες επιχειρήσεις μικρομεσαίες Ιδίως ε, στα ανατολικά κράτη-μέλη, επειδή οι χώρες αυτές, τα μόσποδα κράτη αυτοί, είχαν πολλές οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, έχουν λοιπόν επιπτώσει. Τι κάνουμε λοιπόν. Θεωρούμε ότι τα πολιτικά μας, ε, οι πολιτικές μας επιδιώξεις είναι σημαντικότερες από την καθημερινή οικονομική πραγματικότητα. Το καταλαβαίνουν αυτό οι πολίτες. Το καταλαβαίνει αυτό η κοινή γνώμη. Ξεκινάμε έναν εμπορικό πόλεμο. Αυτό το θέμα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως πολιτική εμπορίου. Ο κύριος Ζαντό. Γιατί μιλάμε, για τη Ρωσία που συμμετέχει και τροφοδοτεί με μια πόλεμο ε, στην Ευρώπη, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είδους κυρώσεις, βέβαια. Το καθεστώς ε, στη Ρωσία σήμερα ελέγχει πλήρως τα μέσα ενημέρωσης ε, και οι κυρώσεις ακριβώς ε, φτιάχνουν ένα οικοδόμημα πολιτικό υποστήριξης του καθεστώτος επιτόπου. Δεν είναι όμως αυτό κάτι το κατάλληλο. Μέχρι τώρα ο στόχος ποιος είναι να αποδομήσουν τη στήριξη στην ολιγαρχία που είναι και διεφθαρμένη γύρω γύρω από τον Πούτιν έτσι. Όταν έχουμε να κάνουμε και φύγουμε κόσμο εκεί από την λιγαρχία αυτή και το αέριο, το πετρέλαιο κλπ που τροφοδοτούν αυτή την κλεπτομανή λιγαρχία και όταν ακουμπάμε οικονομικές πτυχές ακριβώς είμαστε επικεντρωμένοι γύρω από ένα τομέα που δεν είναι ότι δεν έχει σχέση άμεση με τον ρωσικό πληθυσμό αλλά ο στόχος είναι να αλλάξει τη σχεσμό δυνάμεων σε αυτήν την ολιγαρχία γιατί μέσω του ελέγχου με τα μέσα και από το παλιό του δίκτυο της ΚΑΤΖΕΜΠΕ, αυτή τη στιγμή που τα λέγει αυτό, ακριβώς εκείνος πλουτίζει αυτό τον κόσμο, αυτήν την λιγορχία που θέλει και έχει πολύ, πολλά χρήματα. Α, λοιπόν θα πρέπει να δούμε αυτή τη συνοχή της θέσης. Το είπαν και οι συνάδελφοι ε, καλύτερα που ε, διέκοψε, πάγωσε την πώληση των Μιστράλ πάνω σε ένα καθεστώς που επαναλαμβάνουμε τροφοδοτεί, ενισχύει ένα αγώνα, μια μάχη, ένα πόλεμο στην Ευρώπη. Και πάνω, δεν ξεχνάμε και τα πλοία ότι έχουν να κάνουν και με τη Σεβαστούπολη εκεί, έτσι, στην Κρυμαία. Αλλά όταν η Φιλανδία υπογράφει μέσω του Κοινοβουλίου με την ε, εταιρεία τη Ρωσική ε, μια συμφωνία. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Όταν ένα μέρος στην Ευρώπη τον, ε, ανήκουν στην Gazprom ε, η αγωγή, αυτό προκαλεί ένα πολιτικό πρόβλημα. Αυτό λοιπόν ε, στις αγκοινέ ενέργειες θα πρέπει να δούμε πώς, εντάξει, τι θα κάνουν οι κυρώσεις αυτές και μέσω της πολιτικής που ασκείται από την άλλη μεριά δεν θα μειωθούν. Τώρα για τις αντί κυρώσεις τα αντίμετρα. Βέβαια, σίγουρα υπάρχουν τα σταθμιστικά που μπαίνουν στη μέση. Έχουμε γεωργούς που είναι και απογοητευμένοι, χάνουν εισόδημα. Αλλά πέρα από το βραχυπρόθεσμο αυτό που χάνεται, τι γίνεται αργότερα όταν έχουμε 150 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο που δίνουμε στη Ρωσία για το πετρέλαιο και το αέριο εδώ στην δέσμη για την ενέργεια, το 40% αυτής, αυτής της δυνατότητας ε, επένδυσης, ναι, στην Ανατολική Ευρώπη, για την εξοικονόμηση ενεργείας. Ε, εδώ θα πρέπει να δούμε και πώς θα ε, μειώσουμε τις εισαγωγές. Άρα λοιπόν διαρθρωτικά τι γίνεται, πώς θα είμαστε λιγότερο εξαρτημένοι από τη Ρωσία και όταν μιλάμε για αγροτικές εξαγωγές. Και εκεί θα πρέπει διαρθρωτικά να δώσουμε μια απάντηση. Γιατί, γιατί στην Ευρώπη παράγουμε ποιότητα και για την ευρωπαϊκή αγορά πρώτα απ' όλα για να έχουμε αυτή την προστιθεμένη αξία αυτή την υπεροχή παρά να υποκύψουμε στην πίεση, κατά την πίεση της διεθνής αγοράς να έχουμε χαμηλή ποιότητα με λίγη προστιθέμενη αξία και που να εξαρτάται από παρόμοιες επαφές. Ναι, κυρώσεις, αλλά στην εσωτερική μας πολιτική αν θέλουμε να μην εξαρτώμαστε από τη Ρωσία, να θα κάνουμε, να δούμε διαδοτικά τι θα κάνουμε, να μην υπάρχουν τόσο ευαίσθητοι τομείς ε, απέναντι στη Ρωσία. Ευχαριστώ. Very much, Mr. Chairman. Uh, first of all... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα σχόλια τα οποία έγιναν σχετικά με την πολιτική πλευρά. Κοιτάξτε, συζητάμε κυρώσεις και οι κυρώσεις εξορισμού είναι πολιτικής φύσεως, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Ε, ε, είναι ε, η φύση τους να είναι πολιτικές. Να επιστήσω την προσοχή σας σε μία επιστολή που είδαμε από τον πρώην πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ρωσία. Τα λέει πολύ εύγλωτα, το διάβασα στο Financial Times σήμερα. Λέει λοιπόν ότι η πραγματική τραγωδία είναι η ε, παρούσα δυτική πολιτική, δηλαδή η ενουσιακή πολιτική. Ε, ε, χτυπούμε την, την ανάπτυξη της Ρωσίας, υποδαβλίζουμε τον εθνικισμό και στην ουσία δίνουμε λόγο στους, στους Ρώσους οι οποίοι έχουν μια πολιταρχική τάση και στην ουσία δεν προωθούμε καθόλου το σωστό διάλογο. Φοβάμαι ότι οι ενωσιακές, ε, τα ενωσιακά όργανα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν στην ουσία βλέπουν μια θαυμάσια ευκαιρία να βγουν στο προσκήνιο της διεθνούς κοινής χωρίς όμως να βλέπουν ε, ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια σχόλια τώρα σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Έμερσον. Τα πλοία Μιστράλ. Αυτό είναι ένα κλασικό ε, ε, ε, το ε, παράδειγμα του τι κάνει η Γαλλία. Η Γαλλία όμως στην ουσία δεν μπορεί να, η οποία προσυπογράφει τις ενωσιακές πολιτικές, δεν βλέπει καθόλου το εσωτερικό της συμφέρον. Ίσως, ίσως θα πρέπει να μάθουν λίγο και ο Κάμερον και ο Μίλιμπαν και όλοι περί αυτών, αυτούς θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα 10 εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι υποφέρουν κυρίως στην Ευρωζώνη ε, ε, ακριβώς λόγω των ε, οικονομικών πολιτικών που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και, οι κεντρικές τράπεζες κυρώσεις ε, της ε, Ρωσίας λέμε ίσως ε, δημιουργήσουν πρόβλημα στην ανάκαμψη. Μα φυσικά και θα δημιουργήσουν. Και σε ποια ανάκαμψη, στην ανάκαμψη των δικών μας χωρών. Και ο κύριος Έμερσον αναφέρθηκε στη Συμφωνία Σύνδεσης. Ο κύριος Έμερσον φαίνεται ότι δεν δέχεται, δεν θέλει, δεν συμφωνεί με αυτήν την περιστασιακή άρση, καθυστέρηση αυτή της συμφωνία. Αυτό είναι απολύτως προκλητικό είδαμε ότι η συμφωνία με τον Καναδά ε, πήρε πέντε χρόνια και γιατί ε, αλλάζουμε τις ε, συνθήκες σε ένα τέτοιο δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Τελευταίο, καμιά φορά λέμε, αναφερόμαστε σε πολιτικούς, δεν είναι εδώ ο κύριος Μποστινάρου που αναφέρθηκε, αλλά και ο κύριος Έμερσον δούλεψε πολλά χρόνια για ένα think tank ε, και ε, προτείνω ο κύριος Έμερσον όταν ε, αφιψηλού κάνει διάφορες θεωρίες οι οποίες όμως τελικά μπορεί να προκαλέσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στις ζωές πολλών ανθρώπων να το σκέφτεται δύο φορές πριν μιλήσει. Κυρία Λεπένα, χωρίς μικρόφωνο η κυρία Λεπέν δεν ακούν οι διερμηνείς. Ναι, είναι λιγότερο δύσκολο. Οι νέοι συνάδελφοι από το ΕΛΚ, από το ΕΛΚ οι νέοι συνάδελφοι πριν από λίγο, έλεγαν τόσο πολλά που βγαίνουν θετικά, αλλά ξέχασε το Ιράκ. Ήταν πολύ θετικό αυτό το εμπάργο. Νομίζω ένα εκατομμύριο παιδιά που πέθαναν από πείνα και επειδή δεν είχαν και φάρμακα παρά τα όσα ζούμε σαν συνέπειες σήμερα και που είναι και συνέπειες αυτού του εμπάργου. Λοιπόν, να προσέχουμε το θέμα των κυρώσεων. Ναι. Ένα μέρο του πληθυσμού νομίζω στην Ουκρανία είναι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν το δικαίωμα. Και άλλοι όμω είναι υπέρ τη Ρωσία και έχουν το δικαίωμα αυτό. Και για να περιληφθεί στη σφαίρα επιρροή ει βάρο τη Ρωσία, αυτό θα οδηγήσει σε μια καταστροφή. Είμαστε σχεδόν κοντά εκεί. Και όλε κυρώσει, κυρώσει, ξανακυρώσει στη Ρωσία. Κάθε φορά που κλιμακώνεται αυτή η κρίση αλλά αυτή η πολιτική κυρώσεων δεν έφερε κάτι το θετικό στην όλη εξαίρεση καταστάσεως στην Ουκρανία. Αντίθετα, παροτρύνει τη Ρωσία που είναι φυσικός ε, σύμμαχος της Ευρώπης να πάει προς άλλους, προς την Κίνα, ας πούμε προς την Ινδία, προς τη Βραζιλία. Και άρα λοιπόν βλέπουμε τις επιπτώσεις αυτής της στρατηγικής. Με κυρώσεις κατά της Ρωσίας τελικά θα έχουμε ένα ε, εμπάργκο δικό τους στο κρασί, στο κρασί, στα γαλακτοκομικά πηγαίνα, στα κρέατα, στα ψάρια κλπ. Οι μίδια αντιμετωπίζουν πρόβλημα κάτω από πίεση οι αγρότες μας στην Ευρώπη. Υπάρχει λόγω του καθεστώτος των ελεύθερων συναλλαγών που εσείς καθιερώσατε και τώρα είναι αποκομμένη από μια σημαντική επικερδή αγορά. Και άρα λοιπόν αυτές έχουν πακροπόθεσμα τρομερά αρνητικές συνέπειες. Χάνουν 1000 ευρώ το μήνα. Τι είναι, το τους αποζημιώνεται, όχι, το ελάχιστον. 5 δισεκατομμύρια χάθηκε, τόσο πόσο αποζημίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 200 εκατομμύρια, άντε και 125 που πριν από προχθές αποφασίστηκαν. Άρα λοιπόν ε, ε, αυτό και μόνο κάνουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω εδώ. Ναι, βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία. Όλα αυτά μετά από το αντίμετρα της Ρωσίας. Οι γεωργοί, οι γεωργοί που υποφέρουν πραγματικά ε, βλέπουμε ότι καταστρέφουν δημόσια κτίρια, βία, γιατί, γιατί χάνονται, γιατί είναι η σταγόνα το νερό που ξεχυλίζει το ποτήρι με το νερό και ακριβώς ε, εμείς είμαστε οι πέτοι και επίσης όλο ε, και περισσότερες δυσπαστικές θέσεις στη Ρωσία, έτσι, γιατί νομίζουν ότι έτσι αντιστέκονται καλύτερα για το θεωρούν σαν αδικία, μια καταπίεση, μια αδικία. Είναι ανόητη, βλακώδης αυτή η πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Εντυπωσιακά ήταν ορισμένα από αυτά που ακούσαμε, ειδικά τώρα τελευταία. Εν πάση περιπτώσει όμως εξακολουθεί να είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Παρακολούθησε αυτά που είπε ο κύριος Έμερσον στην παρουσίασή του και ορισμένα σημεία ήταν εξαιρετικά σημαντικά. Έχουμε τρεις επιλογές. Η μία επιλογή είναι να μην κάνουμε τίποτα. Και αυτό σημαίνει ότι στην ουσία η Ρωσία αφήνεται να κάνει ό,τι θέλει. Θέλει να πάρει την Ουκρανία, παρακαλώ, περάστε. Θέλετε να πάρετε τη Μολδαβία, παρακαλώ, τη Γεωργία επίσης. Θέλετε να περάσει, θέλει η Ρωσία να περάσει λίγο τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν βαριέσαι, το κάνει. Δεύτερη επιλογή είναι οι ε, ουσιαστικές αποτελεσματικές κυρώσεις. Εδώ από την παρουσίαση του κυρίου Έμερσον ε, προκύπτει ε, και αυτό είναι άσχετο τη συζήτηση για το κατά πόσον εγώ πιστεύω ε, το ότι οι κυρώσει είναι σωστέ ή όχι, ε, ότι δεν είναι πολύ αποτελεσματικέ οι κυρώσει γιατί είναι ελλειπεί, είναι μερικέ και δεν, έχουν, δεν έφτασαν την κατάλληλη ε, στιγμή ενδεχομένω ε, μας είπε ότι θεωρούν παράσημο μερικές φορές ε, οι Ρώσοι αυτές ε, τις ε, ε κυρώσεις. Αυτό μπορούν να το κάνουν γιατί στην ουσία είναι, δεν, είναι, πολλ, δεν είναι πολλές, δεν είναι όσες θα έπρεπε και δεν είναι σε τομείς που πραγματικά να τους δημιουργούν πρόβλημα. Θα έπρεπε και στην, στον αθλητισμό και στο, στο ποδόσφαιρο και σε αυτά θα έπρεπε να έχουμε τέτοιου είδους κυρώσεις κυρώσεις, αλλά ε, θα έπρεπε να ε, παγώσουμε και τους ε, λογαριασμούς όλων αυτών που λένε πω ότι κακιά που είναι η Δύση, αλλά τα παιδιά τους σπουδάσουν στη Δύση και έχουν λογαριασμούς και χρήματα στη Δύση. Εάν θέλουμε δηλαδή πραγματικά να μην περάσουμε στο τρίτο, στον πόλεμο, ή αν θέλουμε πραγματικά αυτές οι κυρώσει να είναι αποτελεσματικές θα πρέπει να τις εφαρμόσουμε με σωστό τρόπο. Εδώ μιλάω για αυτούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπαθούν να μην ε, ε, ε, πάρουν ποινές, να μιλήσουν με λίγο πιο διπλωματικό τρόπο, να συνεχίσουμε δηλαδή τις διπλωματικές συζητήσεις, να μην πάρουμε αποφάσεις για το εμπορίο. Πιστεύουμε ότι αυτοί έχουν μια κρυφή ατζέντα, γιατί αν δεν κάνουμε τίποτα και αφήσουμε τη Ρωσία να παίξει μόνη της, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταρρεύσει και τότε αυτοί οι άνθρωποι ίσως να πετύχουν αυτό που θέλουν αλλά θυμηθείτε, αν αυτό συμβεί, ε, τότε οι αγαπητοί Ρώσοι φίλοι τότε θα έρθουν και θα σας κυνηγήσουν ε, και τότε θα πρέπει και τότε εσπευμένα θα ζητήσετε τη βοήθεια των Αμερικανών. Υπάρχει και μια τέταρτη οδός. Υπάρχει μια τέταρτη οδός της πολιτικής και της διπλωματίας και πρέπει επιτέλους σοβαρά να κάνουμε αυτό που λέει η συνθήκη του Λισαβόνα. Ναι, έχουμε μια κοινή πολιτική εξωτερικών και άμυνα ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τώρα έχουμε 28 διαφορετικέ εξωτερικέ πολιτικέ και πολιτικέ ασφαλεία και αμυντικέ πολιτικέ. Και απέχουμε πολύ από μια κοινή προσέγγιση. Και όταν προκύψει μια σύγκρουση, προσπαθούμε τώρα με ελάχιστα μέσα ε, σαν να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μία αρκούδα με βελόνες. Οι βελόνες πονάνε λίγο αλλά δεν κάνουν τίποτα ιδιαίτερο. Χαίρομαι πολύ που ο κύριος Έμερσον αναφέρθηκε στην περίπτωση του Γεφτουσέγκοφ και την εταιρεία του συστήμα. Βοηθάμε τον Πούτιν στην ουσία να ενισχύσει τη δύναμή του. Δηλαδή, όσα δίκτυα και όσοι ολιγάρχες δεν ήταν ακόμη υποτελείς στην Νέφτ και στην Rosneft και στην Gazprom και την Rosneft υποχρεώνονται και αυτοί να συμμορφωθούν και καταλήτης για την ε, περίπτωση Γεφτουσέγκοφ ήταν η προσπάθεια να αγοράσει μια εταιρεία που λεγόταν Basneft που ήθελε να την αγοράσει και η Rosneft και με ρωσικό τρόπο αντιμετωπίστηκε αυτό και οι μετοχές των εταιριών του Γευτουσεύκο πέφτουν, η τράπεζά του πολίθηκε και ο Πούτιν αυξάνει ακόμη περισσότερο τη δύναμή του. Και ακόμη ε, και στο Ουσμπεκιστάν ε, ε, αυξάνεται η δύναμη των συμμάχων του Πούτιν. Στην ουσία λοιπόν εδρεώνει ακόμη περισσότερο τη δύναμή του. Αντί να αποσταθροποιείται και σε κάποιους τομείς διαπιστώνουμε επιπτώσεις. τα ποσοστά μπορεί να ακούγονται μικρά, αλλά για συγκεκριμένους τομείς μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Και όταν συμβαίνει αυτό που άκουσα ότι κάνουν κάποια κράτη-μέλη, ότι για παράδειγμα υπάρχουν τάσεις προστατευτισμού, ότι δηλαδή κάποιες ε, παραδόσεις εμπορευμάτων για κάποια σούπερ μάρκετ καθυστερούν ε, λόγω γραφειοκρατικών ε, ταλαιπωριών, τότε παραβιάζουμε και τους κανόνες της δικής μας ενιαίας αγοράς. Πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε την κατάσταση με τη Ρωσία, να διευκρινίσουμε ότι αυτά που κάνει με την Ουκρανία δεν είναι σωστά, αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω μιας κοινής πολιτικής αυτή είναι και η συμβατική μας υποχρέωση. Θα πρέπει λοιπόν οι 28 Υπουργοί να το κάνουν. Χαιρόμαστε για τη συμφωνία σύνθεσης με την Ουκρανία, αλλά όπως ανέφερε και ο κύριος Έμερσον, το ελεύθερο εμπόριο που ήταν η ουσία της συμφωνίας, την παγώσαμε. Αυτό το τμήμα το παγώσαμε για 1,5 χρόνο. Δηλαδή πώς εξυπηρετούμε και τους Ουκρανούς με αυτά που κάνουμε. Υπόθηκε ότι ένα τρίτο των υποδομών ενέργειάς μας ανήκει ε, στους ε, Ρώσους. Στην περίπτωση της Γερμανίας ένα δεύτερο τρίτο ανήκει στους Κινέζους και το τρίτο τρίτο ανήκει στην, ε, σε Ευρωπαίους εταίρους. Είναι σωστά αυτά που έχουμε κάνει. Ο κύριος Ομπεμάε τελευταίος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα νέες προσπάθειες ορισμού των ευρωπαϊκών αξιών. Τώρα λέγονται ευρωατλαντικές, ε, ότι είναι ευρωατλαντικές αξίες. Και νομίζω ότι πολλές απόψεις είναι σαν θρησκευτικέ απόψεις. Το σημαντικό είναι αυτό που υπόθηκε από τον ε, επιστήμονα. Είναι σημαντικές οι κυρώσεις αλλά δεν αλλάζουν τίποτα. Είναι σημαντικό να ακούσουμε αργότερα τι επίπτωση θα έχουν. Γιατί δεν είναι αποτελεσματικές αυτές οι κυρώσεις. Αλλά γιατί παρόλα αυτά είναι σημαντικές. Αυτό πρέπει να το πούμε στους ε, εκλογείς μας. Είναι λυπηρό να διαπιστώνουμε ότι, ότι η γεωργοί μας χρειάζεται να καταστρέψουν τα προϊόντα τους. Το διαπιστώνουμε αυτό και στην ε, Γερμανία και στην Αυστρία. Και ήδη υπολογίζουμε ότι θα έχουμε εκατομμύρια απώλειες φέτος. Πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε στους πολίτες μας. Τι στόχο έχουν όλες αυτές οι κυρώσεις, ούτως ώστε ενδεχομένως ή και όχι να τη στηρίξει ο πληθυσμό. Είναι πολύ δύσκολο. Ακούω από κάποιον προλαλήσαντα ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τον πληθυσμό. Αλλά δεν έχουμε, πρέπει να υποστηρίξουμε τους ε, γεωργούς που ε, έκαναν ό,τι μπορούσαν, που έκαναν την ε, συγκομιδή των προϊόντων τους και τώρα δεν μπορούν να τα πωλήσουν. Χάνουν το εισόδημά τους για τις επιτυχείς κυρώσεις. Κάποιοι αναφέρθηκαν στο Ιράν. Πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι υπήρξε κινητικότητα στην περίπτωση του Ιράν έχει να κάνει με γεωστρατηγικούς παράγοντες και την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων Σουνιτών Σιητών. Αλλιώς ε, θα είχαμε διαπιστώσει ότι παρά το ότι είχαμε κυρώσεις επί 30 χρόνια η δυνατότητα αντίστασης ε, μιας κλειστής χώρας είναι μεγάλη. λέγονται ε, ωραία λόγια, αλληλεγγύη, ε, σοβαρότητα, αλλά θα πρέπει να έχουμε και αριθμητικά στοιχεία. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στους δύο εκπροσώπους της Κομισιόν. Πρώτος ο κύριος Κλακ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αναφέρω κάποια στοιχεία και εν πάση θα μιλήσω ε, για, ε, σαν εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης γεωργία. Δεν θα αναφερθώ στο γενικότερο γεωπολιτικό ζήτημα. Ο κύριος Έμερσον είπε ότι δεν θα πρέπει να ε, υπερβάλλουμε αλλά ούτε και να υποτιμούμε το εύρος των κυρώσεων. 10% των ε, γεωργικών μας εξαγωγών ε, κατευθύνονται στην Ρωσία. Ε, και στο εμπάργκο αυτό συμπεριλαμβάνεται περίπου το μισό των 5 δις τα οποία φορούν αυτά τα 10%. Γενικώ έχουν επιλεγεί αυτές οι κυρώσεις οι οποίες θα πονούσαν ιδιαίτερα τις χώρες οι οποίες πρωτοστάτησαν στην λήψη των μέτρων. Ε, και επίσης ε, ε, έχουν φύγει, έχουν βγει από, τις, από τους περιορισμούς αυτά τα προϊόντα τα οποία η ίδια η Ρωσία θέλει να εξακολουθεί να προμηθεύεται. Επίσης γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι ένα 1,5% ε, ε, ε, είναι το ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύεται στο ΑΕΠ. Ε, αυτό βεβαίως, βεβαίως υπάρχουν χώρες οι οποίες πλήγον, πλήττονται ιδιαίτερα, έχουν ιδιαίτερα πληγή ας πούμε ε, σε ορισμένες περιπτώσεις ε, περιοχές οι οποίες είναι της υπαίθρου και οι οποίες ήδη αντιμετώπιζαν προβλήματα ιδιαίτερα ευάλωτες. Προσπαθούμε να λάβουμε μέτρα έτσι ώστε να γίνουν πιο ήπιες οι επιπτώσεις των μέτρων που έχει λάβει η Ρωσία. Ε, ε, συχνά επικρίνεται η κοινή γεωργική πολιτική, ωστόσο πιστεύω ότι και με τις απαντήσει ε, τις οποίες δώσαμε δείξαμε ότι έχουμε την δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε σε τέτοιες επίγουσες καταστάσεις. Πάρα πολύ γρήγορα, ήδη από τον Αύγουστο, βάλαμε κάποια μέτρα επίγοντα έτσι ώστε να στηρίξουμε τον τομέα των, φρύτων, των φρούτων και των λαχανικών που επλήγησαν ιδιαιτέρως Επίσης προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την εξέβρεση εναλλακτικών αγορών για να μην ε, ε, κατακριμνιστεί η αγορά. Όσον αφορά τα γαλακτοκομικά και εδώ ε, βάλαμε κάποια άλλα εργαλεία της ΚΑΠ. Χρησιμοποιήσαμε την ιδιωτική για τη δημόσια αποθήκευση έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα ιδιαίτερα με τις τιμές επαναλαμβάνω ότι και σε αυτή την περίπτωση η ΚΑΠΑ απέδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει, όχι βεβαίως να άρει τις αρνητικές επιπτώσεις, αλλά να βοηθήσει. Μέσω πρόθεσμα τώρα λαμβάνουμε δύο είδη μέτρων προσπαθώντας ε, να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Πρώτον, προσπαθούμε να επιταχύνουμε όσο γίνεται περισσότερο ε, τις διαπραγματεύσεις ελευθέρων, συμφωνιών συγγνώμη, ελευθέρου εμπορίου με διάφορες ε, χώρες ε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να επιτύχει κανείς μια τέτοια συμφωνία FTA δηλαδή εν μια ανοιχτή. προσπαθούμε να κάνουμε πιο γρήγορα. Επίσης προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες, κάποιους επίμονους μη δασμολογικούς φραγμούς. Ας πούμε προχωρήσαμε σε ε, ε, διορθώσεις όσον αφορά την εξαγωγή βοήου κρέατος στην Τουρκία ή φρούτων και λαχανικών εις τις Ηνωμένε Πολιτείε. Επίσης ε, χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή, Πολιτική, μια, η Ευρωπαϊκή Ένωση μια νέα πολιτική προώθησης. Με τον τρόπο αυτό δίνουμε περισσότερη χρηματοδότηση στους γεωργούς έτσι ώστε να στραφούν προς τις εξαγωγές προσπαθώντας να βρουν νέες ε, αγορές. Έχουμε δημιουργήσει ένα νέο ταμείο το, το προηγούμενο μήνα έτσι ώστε να μπορέσει να αντισταθμιστεί ε, το, να αντισταθμιστούν τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει λόγω της, ε, του εμπάργου προς τη Ρωσία. Αυτή η γενικότερη πολιτική προώθηση των προϊόντων πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει στην εξέβρεση εναλλακτικών αγορών εναλλακτικών σε σχέση με την ε, Ρωσία. Και με τον τρόπο αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, ε, προσπαθούμε ε, και, και καταφέρνουμε, αν όχι πλήρως, τουλάχιστον εν μέρη, να εξισορροπήσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Μάρτιν Λούκας, νομική υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα όμως να δώσω το λόγο ε, στον ε, υπεύθυνο για τις δημιουργίες, στην υπεύθυνο για τις διμερείς σχέσεις με τη Ρωσία. Ε, εργάζομαι λοιπόν στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου στο τμήμα σχέσεων με την Ρωσία. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, δύο σε αυτά που ακούστηκαν. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ε, η Ρωσία ε, έβαλε ένα εμπάργο που αφορά περίπου 5 δις ε, ευρώ. 1,4 ε, αφορά το χείριο κρέας, ε, το οποίο όμως το γνωρίζαμε ήδη από τον Ιανουάριο και βεβαίως είναι και θέμα προστατευτισμού της αγοράς. Επίσης, ένα δις ή κάτι παραπάνω αφορά τα αχλάδια με προέλευση Πολωνία. Η Ρωσία παρουσίασε τα ε, μέτρα αυτά ως πολιτικά, αλλά κατά την άποψή μας ε, κρύβουν ε, τον προστατευτισμό τον οποίον ούτως ή άλλως ήθελε να εφαρμόσει ο κύριος Πούτιν έτσι ώστε να δώσει την δυνατότητα στη βιομηχανία της χώρας του να αναπτυχθεί χωρίς εξωτερικό ανταγωνισμό. Πριν από τρία χρόνια ξεκίνησε αυτήν την σειρά προστατευτικών μέτρων η Ρωσία στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ε, εν τω μεταξύ όμως ε, δεν ε, έχει προχωρήσει, δεν έχει προοδεύσει η οικονομία σε αυτούς τους τομείς. Εν πάση περιπτώσει εδώ βλέπω ότι προσπαθείτε να αποτιμήσετε το θετικό ή όχι αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι κυρώσεις. Δεν μπορούμε να, κάνουμε, πούμε πούμε εμείς κάτι. Βεβαίως εμείς ε, ε, σκεφτήκαμε αλλά το Συμβούλιο αποφάσισε τους, ε, τις κυρώσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έμερσον. Thank you very much. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αρκετές ερωτήσεις και ενδιαφέροντα σημεία. Με συγχωρείτε, αλλά από εδώ που κάθομαι δεν βλέπω τα ονόματα. Έχω τη σειρά με την οποία μίλησαν. Βλέπω τον κύριο Ντάκμουθ εδώ, γιατί είναι πολύ κοντά μου, αλλά δεν βλέπω τα υπόλοιπα ονόματα. Λοιπόν, για την πρώτη παρέμβαση, οι ρωσικές τράπεζες. Νομίζω ότι οι ρωσικές τράπεζες υφίστανται σοβαρή ζημιά τώρα και το Κρεμλίνο αμέσως αρνήθηκε να δώσει βοήθεια σε μερικές που το ζήτησαν, αλλά σε τελευταία ανάλυση η κυβέρνηση της Ρωσίας έχει αποθέματα 400 δις δολάρια και δεν θα επιτρέψουν σε μια τράπεζα να ε, πτωχεύσει, θα τις διασώσουν για τον τομέα του πετρελαίου. Ναι, τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να καθυστερήσουν σοβαρά την βελτίωση και την επέκταση του πετρελαϊκού κλάδου γιατί πρέπει να ανοίξουν και νέα ε, νέα πεδία άντλησης πετρελαίου. Αλλά αυτό είναι μακροπρόθεσμο και η κρίση στην Ουκρανία μπορεί να κλείσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί αν επιτύχουμε αυτά που θέλουμε για την Ουκρανία, σε λίγο θα επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση αλλά για το φυσικό αέριο. Δεν έχει αναφερθεί ακόμη. Δεν έχει ρόλο ακόμη το φυσικό αέριο. Γιατί αν σταματήσει η Ένωση να, αγοράσει, να αγοράζει φυσικό αέριο από τη Ρωσία, θα έχει μεγάλο ρόλο στα σοβιτικά έσοδα. Αλλά βεβαίως έχουμε πολλά αποθέματα φυσικού αερίου. Για μερικούς μήνες θα μπορούσαμε χωρίς ε, εισαγωγές από πλευράς τους. Από σήμερα όμως η αγωγή δεν είναι παρκώς πλήρης και η άλλη υποδομή. Εμείς ε, ζητήσαμε κάποιες υποδομές, έναν ε, κατάλογο νέων εγκαταστάσεων για τη μεταφορά του αερίου, αλλά δεν θα τον έχουμε, δεν θα έχουμε αυτές τις αναγκαίες υποδομές πριν το 2020. Εάν λοιπόν η Ρωσία θεωρήσει ότι θα πέσουν απότομα τα έσοδά τους από το φυσικό αέριο θα τους ανησυχούσε ιδιαιτέρως αλλά θα πάρει χρόνο αυτό και οι διπλωμάτες μας ε, που μιλούν από πλευράς της Gazprom μπορούν να δημιουργήσουν αρκετή σύγχυση για να μην συμβεί. Δεύτερον, ο δεύτερη, η δεύτερη παρέμβαση, αποτελεσματικότητα των κυρώσεων. Τι πραγματικά επιδιώκουμε σε σχέση με την Κρυμαία. Ε, τώρα ε, μιλάω εξ ονόματός μου και μόνο. Η δική μου ερμηνεία των στόχων της Ένωσης είναι η Ρωσία να φύγει από την Ουκρανία. Να επιτρέψει στην Ουκρανία να αποφασίσει για τη μοίρα της. Αυτός είναι ο στόχος, όχι τι συμβαίνει. Μια δεύτερη ερμηνεία μου για την Κρυμαία και ένα διπλωμάτη σίγουρα δεν θα το έλεγε θα ήταν εάν ο Πούτιν μετά την προσάρτηση της Ουκρανίας είχε πει σταματάω εδώ και θα είμαι απόλυτα συνεργάσιμος ε, σε σχέση με την Ουκρανία υποθέτω ότι οι ηγέτες μας θα είχαν πει εντάξει, οκ, okay, ας συμφωνήσουμε αλλά δεν συνέβη γιατί η Ρωσία επετέθη και ε, εισβάλλει όλο και βαθύτερα στην Ουκρανία. Ήμουνα σε μια σημαντική διάσκεψη στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα και θεωρώ ότι το χειμώνα θα ξαναπροκύψει πρόβλημα Κρυμαίας. Δηλαδή, θα είναι δύσκολη η κατάσταση της Κρυμαίας από πλευράς ίδρευσης, ε, ηλεκτροδότησης και η Ρωσία πρέπει να έχει μια χερσαία δίωδο προς την Κρυμαία μέσω της Μαριούπολης και πέραν της Μαριούπολης Άρα πολλοί στο Κίεβο περιμένουν ότι μετά από μια περίοδο ύφεση νέα επίθεση για να υπάρξει χερσαίος διάδρομος ε, Ρωσίας Κρυμαίας. Λοιπόν να το περιμένετε αυτό. Τρίτον. Τρίτη παρέμβαση. Έθεσε θέματα των ε, αμυντικών δυνατοτήτων. Σας παρακαλώ να συνδέσετε μερικές ερωτήσεις ε, για να συντομεύουμε. Παρακαλώ ορισμένες ερωτήσεις να τις απαντάτε από κοινού. Λοιπόν, για τις αμυντικές δυνατότητες. Εγώ είμαι ναι. Επόμενη ερώτηση. Εγώ από πλευρά μου προσωπικά λέω ναι, βεβαίω. Διάφορα θέματα για τη γεωργία. Βεβαίω να αναθεωρήσω το κείμενό μου και να μειώσω στο μισό τις γεωργικές εξαγωγές που θίγονται αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμη μικρότερες επιπτώσεις από ότι αυτές που αναφέρω εγώ στην εργασία μου. Για τους στόχους αναφέρθηκα. Νομίζω ότι οι στόχοι μας είναι να μπορεί η Ουκρανία να δράσει ανεξάρτητα και ένας ε, λίγο πιο ασαφής, ε, πιο μακροπρόθεσμος στόχος να βοηθήσουμε να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη Ρωσία, αλλά αυτό είναι μακροπρόθεσμος στόχος, ε, μεγαλόπνος, απέχουμε πολύ. Τώρα, εάν στόχος μας είναι να απογοητευτούν τόσο πολλοί οι ολιγάρχες που να πιέσουν το Κρεμλίνο να αλλάξει πολιτική, ναι, να το συζητήσουμε, αλλά δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό. Οι ολιγάρχες χρειάζονται στήριξη οικονομική από το Κρεμλίνο και θα συνεχίσουν να τη χρειάζονται. Άρα δεν το περιμένω αυτό. Αντίμετρα τώρα εάν η Ένωση πραγματικά μείωνε πάρα πολύ το φυσικό αέριο που εισάγει θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίμετρα για παράδειγμα την απαλωτρίωση των συμφερόντων της Total και της BP Τώρα για αυτά που είπε ο κύριος Ντάρτμουθ. Λόρδος Ντάρτμουθ λέγομαι. Λέει ο κύριος Ντάρτμουθ. Έχουμε... Έχω πολύ διαφορετική προσέγγιση για το ποιος προκαλεί ποιον. Ως οικονομολόγος ο πρέπει να πω ότι ο Πούτιν αποφάσισε ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να μπει σε τελειονιακή ένωση με τη Ρωσία, αλλιώ θα τη επιτέθετο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε πάντα ότι θέλουμε ενό υψηλού επίπεδου συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Ουκρανία, αλλά θα θέλαμε και η Ρωσία να έχει, συγγνώμη να έχει μια συμφωνία εμπορίου με τη Ρωσία και άλλες χώρες θεωρούμε ότι όπως και η Μολδαβία και η Γεωργία θα θέλαμε να, έχουμε, να έχουν καλές εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία. Αλλά ο Πούτιν είπε όχι. Εγώ τα θέλω όλα και μόνο εγώ. Δεν συμφωνώ λοιπόν ότι η συμφωνία σύνδεσης ε, ήταν πρόκληση για τη Ρωσία. Για τη Γεωργία τα είπαμε ήδη. Περαιτέρω κυρώσεις ποδόσφαιρο, παγκόσμιο κύπελο. Ναι, καλή ιδέα. Τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό. Τελείως ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Έμεσον. Νομίζω ότι συζητήσαμε ουσιώδεις πλευρές, δηλαδή και τις επιπτώσεις για τη Ρωσία, αλλά και τις επιπτώσεις για την Ένωση των Αντιμέτρων. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και τα δύο αυτά θέματα. Αυτή η ζήτηση θα συνεχιστεί οπωσδήποτε. Και κυρίως ε, θα συνεχίσουμε να ασχολούμεθα με τα θέματα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Σημείο 13. Ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση τον ΙΠΑΣ. Εδώ και 12 χρόνια έχουμε διαπραγματεύσεις για το ΙΠΑΣ. Για πολύ καιρό δεν ε, υπήρξαν πολλές εξελίξεις. Τον περασμένο μήνα υπήρξε κάποια κίνηση και πρέπει να το συζητήσουμε λίγο περαιτέρω. Χαίρομαι που είναι εδώ η Σάντρα Γκαλίνα που ασκεί καθήκοντα διευθυντού και είναι ματάρχης Είπα στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου παρακαλώ να μας πείτε τι γίνεται πώς έχουν τα πράγματα και τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων είπα και το θέμα της χρονικής εξέλιξης και το θέμα της εφαρμογής τους Σας δίνω το λόγο. καλύτερες ευχές μου για την ε, νέα σας θητεία. Πρώτη φορά έρχομαι ενώπιόν σας. Ελπίζω να έχουμε τόσο καλές ε, σχέσεις όπως και στο παρελθόν. Ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να σας παρουσιάσω την κατάσταση για τις ε, οικονομικές, για τις συμφωνίες οικονομικών εταιρικών σχέσεων, EPAs. Καλό είναι λοιπόν να έχετε μια συνολική άποψη. Όπως τα ξέρετε, καταλήξαμε τις διαπραγματεύσεις EPA με δύο αρκετά μεγάλες περιοχές, Δυτική Αφρική και είμαστε σε διαπραγματεύσεις με την περιοχή EAC. Μια σειρά από χώρες όπως το Καμερούν και το Φίτζι έχουν επικυρώσει και περνάνε τώρα στην εφαρμογή. Θα την εφαρμογή και μετά να μιλήσω για τις υποδιαπραγμάτευσεις συμφωνίες. Εφαρμόζουμε λοιπόν πλήρως την EPA, την συνολική EPA για την Καραϊβική. Έχουμε ενδιάμεσες EPA με την Παπουασία Νέα Γουζέα, Γουινέα Φίτζι, το Φίτζι, τα Φίτζι, με την περιοχή της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής Ζιμπάμπουε, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος και Σεϊχέλας, και τώρα ξεκινάμε την εφαρμογή με το Καμερούν και την Καραϊβική. Υπάρχει πρόοδος. Η συμφωνία αυτή ε, εφαρμόζεται προσωρινά εδώ και χρόνια. Ορισμένες χώρες και από την πλευρά μας ολοκληρώνουν τη διαδικασία επικύρωσης. Έχουμε τακτικές συναντήσεις η επόμενη συνάντηση για θέματα εμπορίου και περιβάλλοντος θα γίνει 18 και 19 Νοεμβρίου. Αν όλα πάνε καλά, η Συμβουλευτική Επιτροπή που είναι ένα από τα όργανα που πρέπει να αναπτυχθεί, να ανθίσει μέσα από αυτές τις EPA, θα έχει συνεδριάσει πριν από την ε, προαναφερθή σας συνάντηση. Δεν σας κρύβω όμως ότι οι τελευταίες μου πληροφορίες μοιάζουν να σημαίνουν δεν θα συμβεί αυτό. Στόχος μας όμως είναι να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Δεν είναι κάτι που εξαρτάται από την Κομισιόν, η Συμβουλευτική Επιτροπή αυτή είναι στα πλαίσια της ΟΚΕ και η κοινοβουλευτική συνέλευση είναι φυσικά υπόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απλώς ενημερωνόμεθα για το τι συμβαίνει. Τι είναι σημαντικό για το Carrefour, για την Καρεβική. Κάναμε μια ανασκόπηση, όπως είχαμε υποχρέωση. Το Carrefour εκπροσωπείται στη Μόνιμη Επιτροπή. Συνεργαζόμεθα πολύ καλά. Έχουμε ένα σύμβουλο που είναι από την περιοχή εκεί. Κάτι σημαίνει αυτό για τους εταίρους μας. Η μελέτη που κάναμε λοιπόν αποδεικνύει ότι θα ήταν πολύ χειρότερη κατάσταση χωρίς μια τέτοια συμφωνία EPA. Τα αποτελέσματα που έχουμε τώρα μπορεί να μην είναι όσα αναμέναμε, αλλά το EPA αυτό, αυτή η συμφωνία, βοήθησε να προστατευτούν οι χώρες κατά την κρίση. Και στον ειρηνικό έχουμε περάσει στην εφαρμογή, πάει αρκετά καλά, συναντώμεθα μια φορά το χρόνο από τότε που αρχίσαμε το 2011 Προηγουμένως συμμετείχε μόνο η Παποσία Νέα Γουινέα, τώρα θα έρθει στην επόμενη συνάντησή μας και το κράτος των Φίτζι. Δεν έχουμε καθορίσει την ημερομηνία, ελπίζουμε να γίνει πριν το τέλος του χρόνου, αλλά δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Θα έλεγα ότι τα αποτελέσματα στην Παπόσια Νέα Γουινέα είναι πολύ εθαρρυντικά. Οπότε διαπιστώσαμε επενδύσεις στην αλληλεία που δεν θα είχαν προκύψει χωρίς το EPA που έχουμε. Ένα EPA εφαρμόστηκε στην Ανατολική και Νότια Αφρική. Είναι η περιοχή των τεσσάρων χωρών που προανέφερα. Έχουμε συναντηθεί με τις χώρες αυτές κάθε χρόνο. Η Επιτροπή έχει συναντηθεί λοιπόν τακτικά. Η επόμενη θα γίνει στο Ζιμπάμπουε. Θέλαμε να γίνει το Νοέμβριο, αλλά από ό,τι φαίνεται συμπίπτει με την μεικτή κοινοβουλευτική συνέλευση. Θα δούμε αν θα γίνει πριν το τέλος του χρόνου ή, θα, ή αν θα πρέπει να αναβληθεί. Λίγα έχω να πω για το Καμερούν. Είμαστε στα πρώτα βήματα της εφαρμογής να συστήσουμε μια επιτροπή, να δούμε τους ε, διαδικαστικούς κανόνες κτλ. Οι συμφωνίες EPA είναι μακρόπνοες. Δεν είναι στόχος αλλά διαδικασία και πολύ σημαντικό είναι ότι είναι εταιρικέ σχέσεις, κυρίως όταν περνάμε στην εφαρμογή. Οι συμφωνίες αυτές χρειάζονται και στο εσωτερικό των χωρών αυτών πολλές μεταρρυθμίσεις. Θέλουμε να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν προς όφελός τους, προς όφελος ε, των επιχειρήσεών τους. Σας καλώ λοιπόν να στηρίξουμε αυτούς μας τους εταίρους. Η Ένωση πρέπει να τους στηρίξει, γιατί οι προκλήσεις, ξέρετε, είναι μεγάλες για πολλές από αυτές τις χώρες. Κάνω λοιπόν έκκληση για αναπτυξιακή βοήθεια. Γιατί για ορισμένες τέτοιες χρηματοδοτήσεις μπορείτε να παίξετε αποφασιστικό ρόλο. Για τις ολοκληρωμένες διαπραγματεύσεις, ολοκληρωθήσεις διαπραγματεύσεις, κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις μας με τη Δυτική Αφρική αρχές του χρόνου, αλλά μετά χρειαστήκαμε κάποιο χρόνο για να έχουμε την μονογράφηση, γιατί μονογραφήσαμε το νομικά ελεγμένο κείμενο. Ήταν μια πολύ επικοδομητική διαδικασία. Εξέφρασαν σαφώς βούληση για να προχωρήσει η κατάσταση οι πλευρές και ελπίζουμε να έχουμε την υπογραφή τάχιστα. Ελπίζω πριν το τέλος του χρόνου. Για την περιοχή Σάντοκ. Έχουμε την Ιγυρία στη Δική Αφρική στο Σάντοκ. Έχουμε μια χώρα μπρικ Μια χώρα BRICS που είναι η Νότια Αφρική. Καταλήξαμε, μονογραφήσαμε ένα μη ελεγχθέν κείμενο, τώρα γίνεται ο νομικός έλεγχος. Η διαδικασία αυτή θα είναι λίγο πιο εργόδης γιατί έχουμε πολλές ε, ε ρήτρες διαφύλαξης ε, και άλλες ε, που χαιρόμαστε που τις επιτύχαμε. Αν δείτε τι έχουμε κάνει, έχουμε 12 λιγότερο αμπτυγημένες χώρες στη Δυτική Αφρική και δύο αλλού που αποφάσαν να μπουν σε EPA αυτό πρέπει να το τονίσουμε, είναι σημαντική επιτυχία. Ήταν πεπισμένοι ότι οι μονομερείς προτιμήσεις ε, δεν θα τους απέφεραν όσο θα τους αποφέρει μια συμφωνία μια συμφωνία EPA. Θέλουν λοιπόν να είναι τμήμα μιας πολυμερούς συμφωνίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλουν επίσης ασφάλεια και σταθερότητα για τις επιχειρήσεις τους γιατί εάν ε, ε, αναπτυχθούν λίγο θα μπουν σε καθεστώς άλλης ομάδας χωρών. Άρα θέλουν να διατηρήσουν το καθεστώς λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Θα πρέπει να τις βοηθήσουμε με ε, μέτρα για ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους. Για τη βοήθεια, βεβαίως, κάνουμε διαπραγματεύσεις με το EAC οι τελευταίες εξελίξεις δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικές δείξαμε όλοι μας την ε, ευλογησία αλλά αυτή η περιοχή τελικά δεν ανταποκρίθηκε στην καλή μας βούληση δεν προσέγγισε τις απόψεις μας σε πολύ σημαντικά θέματα όπως ε, το άρθρο για τη μη εφαρμογή που είναι αντιγραφή του άρθρου 96. Δεν ξέρω αν σας κούρασα. Ευχαριστώ που μας καλέσατε να σταματήσω εδώ αν έχετε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ, David Martin. Ευχαριστούμε. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω ως άντρα στην Επιτροπή. Είχαμε καιρό να τα πούμε και χαίρομαι γιατί ακούω και για καταστάσεις οι οποίες έχουν προχωρήσει και αυτό είναι καλό. Λυπούμε και εγώ που η Κοινή Συμβουλευτική Επιτροπή δεν είναι ακόμα σε επιχειρησιακό επίπεδο, δεν λειτουργεί. Ε, είπες ε, ότι δεν ε, είναι ευθύνη της, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά η και με, πίεζε και μένα προσπαθούσε να μου πει ότι στην ουσία δεν είναι ούτε δικιά τους ευθύνη και επομένως ίσως θα πρέπει να διευθετηθεί το θέμα οργανωτικά. Όσον αφορά τα Φίτζι και εγώ χαίρομαι που υπάρχει μια συμφωνία που βρίσκεται στα σκαριά ε, αλλά θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει το λεγόμενο sugar money για τα Fiji. Ε, το οποίο δεν θα βοηθούσε ενδεχομένως τα ίδια Φίτζη αλλά ορισμένες, ε, ε, ορισμένες την ευρωπαϊκή πλευρά κυρίως ορισμένες εταιρείε οι οποίες πολύ θα ήθελαν απελευθέρωση αυτών των sugar money επίσης Αναρωτιέμαι τώρα που εντάσσονται τα Φίτζι σε αυτές τις συμφωνίες ε, τι θα γίνει με τα LDC στην Αφρική αν μπορούμε δηλαδή ε, να φτάσουμε ε, σε ένα ικανοποιητικότερο επίπεδο συμφωνιών γιατί εκεί είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλό το επίπεδο μπορεί να γίνει δηλαδή ένα περιφερειακό πλαίσιο Δυτική Αφρική Ομολογώ ότι δεν το κοίταξα από πολύ κοντά, δεν το τσεκάρισα, αλλά ε, συνδικάτα μου λένε ε, ότι οι εργασιακές ε, ρήτρε δεν είναι σωστές όσον αφορά την Economic Partnership Agreement με την Δυτική Αφρική. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην ε, ε, βιομηχανία των φοινικόδεντρων ε, και θα πρέπει να δούμε λίγο το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων εκεί. Επίσης, συγχαρητήρια σχετικά με το θέμα αυτό των γεωγραφικών ενδείξεων για τα γεωργικά προϊόντα. Ήταν μια καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Um, for your uh, Ευχαριστώ. Σύντομες ερωτήσεις. Δύο συγκεκριμένα. Ε, πρώτον, υπάρχει σχετικός προβληματισμός ε, έστω και αν ε, οι αρχικές προθέσεις των διαπραγματευτών για για, τους, ε, για τη συμμετοχή των εκπροσώπων από την Αφρικανική Ένωση. Ε, ποιος είναι ο προβληματισμός τους, ε, υπάρχει κάποια παρανόηση, νομίζω ότι είναι ε, καλό να υπάρχει καλή πίστη από όλους τους εμπλεκόμενους σε μια διαπραγμάτευση και πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Δεύτερον, όσον αφορά την αιρεσιμότητα, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει ήδη κάποιο προσχέδιο, πώς ε, έχετε κάποιες πληροφορίες να μας πείτε όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Η Λόλα νομίζω έχει ζητήσει πρώτα το λόγο και μετά εγώ λέω κύριο Σόλτς. Α, να μιλήσω εγώ, ωραία. Κανένα πρόβλημα. Η ΕΣΥ, η Κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής, Η κυβέρνηση της Ναμίμπια χαιρέτησε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Είπαν ότι χαίρονται που καταργήθηκαν οι δασμοί για τα, για τα προϊόντα τους και τις εξαγωγές πρώτων υλών. Ισχύει αυτό. Γιατί Εάν το κατάφερε αυτό η Ναμίμπια δεν μπορεί να γίνει και στη συμφωνία με την Ανατολική Αφρική κάτι παρόμοιο. Γιατί νομίζω ότι προκαλεί πολλές ε, δυσχέρειες. Ε, τις δυσχέρειες που προκαλεί και η ρήτρα για τη μη εφαρμογή. Είπατε ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Ανατολική Αφρική, αλλά χτες στον κενιανικό τύπο αναφέρθηκε ότι έχουν κλείσει οι διαπραγματεύσεις. Κατέληξαν. Τι ισχύει. Ολοκληρώθηκαν. Οι διαπραγματεύσει θα υπάρξει κατεξοδότηση πράξη ε, για την εφαρμογή. Και η Δυτική Αφρική είπατε ότι θέλετε να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών και να υπάρχει διαφάνεια. Νομίζω ότι ίσως ε, έχουν παίξει ρόλο κάποιες υψηλότερες δυνάμεις ε, που δεν μας εκπλήσει εμάς αλλά εκπλήσει την κοινωνία των πολιτών σε αυτήν την περιοχή και γι' αυτό υπάρχουν και διαμαρτυρίες στην κοινωνία των πολιτών. Παρενέβησαν λοιπόν κάποιες τέτοιες ε, δυνάμεις για να υπάρξει κατάληξη. Πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό. Σκά. Ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε αυτές τις τελευταίες πληροφορίες. Έχω μια ερώτηση όσον αφορά τα νησιά Φίτζι. Προβληματίζομαι λίγο για την προσέγγιση. Ε, όταν αποφασίστηκε και αποφάσισε το Συμβούλιο ε, ε, να ασκήσει κυρώσεις μετά από το πραξικόπημα ε, βλέπουμε να προωθείται η EPA. Μπορείτε λίγο να μας διευκρινίσετε την κατάσταση και επίσης με ποιο τρόπο ας ερμηνεύεται η δέσμευση των, των της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, We heard from Τις χώρες ε, ECOWAS. Εκεί ξεκίνησε το EPA τον Ιούλιο. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα μέλη της περιοχής αυτής ε, θα έχουν ακριβώς το ίδιο καθεστώς από την 1η Οκτωβρίου. Ε, ναι, αλλά φαίνεται ότι η κατάσταση στην Κάνα, στην ακτή του ε, ε Ελεφαντοστού κλπ. Ε, έχουν διαφορετική προσέγγιση γιατί φαίνεται ότι εκεί ισχύει το ενισχυμένο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και βλέπουμε ε, μάλιστα εκεί να υπάρχει και κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την περιφερειακή ε, ολοκλήρωση αλλά και την πρόσβαση στην αγορά. Έχουμε το άρθρο 2 του κανονισμού για την πρόσβαση στην αγορά που λέει ότι που λέει ότι η Κομισιόν θα τροποποιήσει το παράρτημα 1 μέσω κατεξουσιοδότηση πράξη σε σχέση ε, με το άρθρο 24α ε, ε, όπως ισχύει στις συμφωνίες με τις χώρες αυτής της περιοχής όπου όμως θα πρέπει να διασφαλίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις του άρθρου κλπ. Ε, μήπως μπορείτε λίγο να μας διευκρινίσετε την κατάσταση κυρίω όσον αφορά αυτή, αυτό το παράρτημα 1 και γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις για την ίδια περιοχή και για το ίδιο EPA. Επίσης, είναι σημαντικό να, πούμε, να μάθουμε ποια είναι τα στάδια της επικύρωσης των διαφόρων EPAs. Ε, γιατί έχουμε συζητήσει πολύ το ε, θέμα του κατά πόσον θα είναι μεικτή συμφωνία αυτή η συμφωνία με τον ε, Καναδά και πρέπει να ξέρουμε λοιπόν και υπό το φως αυτό ποιοι θα επικυρώσουν τις EPA. Ε, Δυτική Αφρική ενδεχομένως ε, λέμε, αναφέρεται ότι θα υπάρχει δυνατότητα ορισμένες χώρες ε, να προστατέψουν μέσω ειδεξιδικευμένων μέτρων την γεωργία τους. Τι θα γίνει όμως το θέμα των καταψυγμένων κοτόπουλων. Δηλαδή, πώς πώς ας πούμε θα αποδείξουν ε, ε, οι παραγωγοί που θα μπουν σε αυτές τις ποσοστώσεις ότι είχαν προβλήματα και τα λοιπά. Ευχαριστώ. Επειδή έθεσαν ήδη ε, ερωτήσεις σχετικά με την κοινωνία των πολιτών, ακούμε τρομερά πολλές σχετικά με την κοινότητα των πολιτών και την ευρωπαϊκή και την αφρικανική. Ακριβώς πέστε μου σας παρακαλώ αυτές οι απαιτήσει σε αυτά τα θέματα πώς λαμβάνονται υπόψη γιατί μερικές φορές υπάρχει έλλειμμα διακυβέρνησης σε ορισμένε εταιρικέ χώρες και εκεί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η κοινωνία πολιτών σε αυτόν τον έλεγχο που μπορεί να ασκείται ακριβώς πώς εδώ αυτό γίνεται και πώς οι παρατηρήσεις σχετικές έχουν ενταχθεί. η Ιλώνα. Σάντσες. Για μας ε, απαράδεκτο είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκβιάζεται τις χώρες ΑΚΕ για να προσυπογράψουν αυτές τις EPA ε, έτσι, και για την συνεργασία, ε, για την ανάπτυξη, την το προσημιακό καθεστώς και εδώ στις αναπτυσσόμενες χώρες όπως και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια δεξάγουμε μια εκστρατεία γιατί πάρα πολλές συμφωνίες γίνονται και είναι συμφωνίες που είναι μειωτικές προς τις χώρες αυτές ε, τις αναπτυσσόμενες. Οι συμφωνίες αυτές που λέγονται ΕΠΑΣ ε, είναι ουσιαστικά ελεύθερων συναλλαγών ε, μασκαρεμένων ε, και κανονικά το ελεύθερο εμπόριο είναι για όλους. Αλλά αυτό δεν υπάρχει καμία ανάλυση θεωρητική, ούτε ιστορική, ούτε εμπειρική, ούτε τίποτα που να το αποδεικνύει. Και υπάρχουν εμποδίζουν την, ε, να προχωρήσουν αυτές τις χώρες και πολλά από αυτά υπάρχει η ρήτρα αναθεώρησης ανοίγει ουσιαστικά την πόρτα για να προχωρήσει κανείς περισσότερο σε αυτές τις ε, επενδύσεις ε, με όλες αυτές τις ζημιές που σημαίνει για, τις, για τον πολιτών σε αυτές τις χώρες που προσυπογράφουν και κάτι ακόμα που ε, υπόθηκε προηγουμένως. Ε, εδώ το 208 παραβιάζεται το άρθρο της Συνθήκης της Αβώνας ε, σχετικά με, τις, με την ανάπτυξη και υποβοηθείται ουσιαστικά η φτώχεια. Και εμείς ε, βγάζουμε το σκαλί που οδηγεί προς την ανάπτυξη ε, Εκείνο όμω δεν του ενδιαφέρει το τι γίνεται αυτό. Και θα ήθελα να ρωτήσω τα δύο πράγματα εξή. Γιατί δεν ακούτε την κοινωνία των πολιτών, όπως το είπαμε και ορισμένα από τα μέλη εδώ. Θα ήθελα επίση να ρωτήσω κάτι για το IT. Τι γίνεται για το ΕΠΑ στο Κάλι Forum. Εδώ ξέρουμε τι συνέπειες θα έχει αυτό. Ευχαριστώ. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση που σχετίζεται με αυτά που είπε και ο Ντέβιν Μάρτιν για τη συμφωνία με τη Δυτική Αφρική. Η Δυτική Αφρική είναι πολύ σημαντική για την παραγωγή κακάο. Ένα μεγάλο τμήμα από τον εισαγωγή μας ε, κακάο έρχεται από την Γκάνα και την ακτή του και ξέρουμε εδώ και καιρό ότι στον τομέα αυτό υπάρχει υποχρεωτική εργασία, ε, παιδική εργασία και εμπορία παιδιών. Το 2012 τα είπαμε αυτά όταν υπήρξε η ένταξή μας στην Συμφωνία για το Κακάο και είπαμε σαφώς ότι θα πρέπει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, να υπάρχουν σαφείς κανόνες για να τηρούνται οι δύο σχετικές συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Και David, κοίταξα το κεφάλαιο βιωσιμότητας στην EPA με τη Δυτική Αφρική. Είναι μισή σελίδα. Χωρίς κανέ, καμία συγκεκριμένη αναφορά που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσει του Κοινοβουλίου. Και ειλικρινά, όταν ε, το διάβασα αυτό είπα δεν μπορώ να δεχτώ έτσι αυτήν την ΕΠΑ. Θα πρέπει να δούμε πώς θα συντάξουμε ένα νοδικό χάρτη που να μας επιτρέψει να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουν σεβαστά αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εάν δεν γίνει αυτό δεν μπορούμε να υπογράψουμε μια τέτοια συμφωνία. Να ξεκινήσω με την ερώτηση του κυρίου Μάρτιν και θα προσπαθήσω να ομοδοποιήσω ε, απαντήσεις ακολουθώντας και τη σειρά των ερωτήσεων ε, θα αναφερθώ και στην κοινωνία των πολιτών και τι προσπαθούμε να πετύχουμε μέσω ε, των EPA για την κοινωνία των πολιτών. Η Συμβουλευτική Επιτροπή ε, κοιτάξτε, ε, ε, εγώ από το 2008 ε, προσπαθώ να επαναλάβω, μάλλον προσπαθούσα να επαναλάβω κάποια, κάποιες προσπάθειες. Εν πάση περιπτώσει τώρα τα καταφέρνουμε από ό,τι φαίνεται. Ε, κοιτάξτε, υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες αφορούν και την κοινωνία των πολιτών. Μία εκ των οποίων είναι ότι έχουμε καλές δομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η ΕΟ και έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη δικιά μας πλευρά, αλλά από την άλλη πλευρά είναι δύσκολο να βρει κανείς έναν ομόλογο ε, οργανισμό ή θεσμό. Ε, ε, και ε, βεβαίως έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αλλά θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να διευθετήσουμε τα τεχνικά ζητήματα πόσα μέλη, γιατί δεν μπορεί να είναι όλα τα μέλη, ποιοι θα έχουν έδρα κτλ. Και ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία να ενταχθούν ακόμα και τα Ελλάς ε, ελάσσονο σημασία, οι ελάσσονε σημασία αναφορέ όσον αφορά ρήτρε για την κοινωνία των πολιτών, οι ρήτρε για οικονομικέ ε, και κοινωνικέ επιτροπέ. Εμεί προσπαθούμε ε, να βρούμε μέσα έτσι ώστε να διευθετηθεί, αυτό που με το ζήτημα τη κοινωνία των πολιτών. Έχουμε τακτικά επαφές και συνεδριάσεις και όπου και οι ε, πρέσβεις ε, παραπονιούνται ε, από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι πολλές φορές παραπονιούνται και για τις συνεδριάσεις PNG. Εν πάση περιπτώσει ε, για την Παπουασία την ε, και Νέα Γουινέα πολλές φορές έχουμε τέτοιου είδους ε, προβλήματα εγώ μπορώ να πω ότι χρειαζόμαστε την κοινωνία των πολιτών και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσω των συμφωνιών αυτών των EPA είναι να εμπλέξουμε και την κοινωνία των πολιτών όσον αφορά δε τα συνδικάτα των χωρών της Ανατολικής Δυτικής συγγνώμη, Αφρικής τους έχω συναντήσει και ε, πραγματικά ε, είναι, θα ήταν πολύ σημαντικό να ακουστεί και η φωνή τους ε, και εδώ γιατί δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να εκφράζονται. Όσον αφορά το κακάο, ασχοληθήκαμε και με το κακάο αλλά βεβαίως δεν ήθελα να ξεσκεπάσω κατά κάποιο τρόπο κανέναν συγκεκριμένα στην συνεδρίαση αλλά πραγματικά δεν θέλω να παίζω με κακούς όρους ε, και δεν θέλω να δείχνω το δάχτυλο σε κανέναν, αλλά... Ε, οι συνθήκες στην Δυτική Αφρική είναι διαφορετικές και άκουσα πολλές αφηγήσει και από πλευρά των συνδικάτων τη Δυτική Αφρικής που μου λένε ότι όλα τα χρόνια έτσι ήταν η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει είναι γεγονό ότι η Δυτική Αφρική ε, βλέπει με πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη, καχυποψία μάλλον θα ε, πω, οπωσδήποτε όλα αυτά τα θέματα. Ε, και ξέρετε ακόμα και αν ε, δεν είναι ε, τυποποιημένη αυτή η συζήτηση έρχεται ο κόσμος και μου λέει τα προβλήματα τα οποία ε, έχουν ακόμα και για την ΑΕΤ μου λένε ότι αν υπήρχε ας πούμε και εγώ από τη δική μου πλευρά αν είχα αυτή την συμφωνία την Economic Partnership Agreement θα μπορούσα διαφορετικά να μιλήσω με την κυβέρνηση της ΑΕΤ Σημερίζομαι την άποψή σας κύριε Πρόεδρε και εγώ, και εγώ ταυτίζομαι πάρα πολύ με αυτήν την κατάσταση και δυσκολεύομαι να την ε, ε, δεχτώ και μάλιστα σε μία ε, περίπτωση απείλησα ότι θα εγκαταλείψω την αίθουσα και είπα ότι εγώ θα φύγω, θα βγω και θα, θα, θα φωνάξω τι γίνεται εδώ μέσα και τι λέτε. Αλλά και για, ε, για, τη Δυτική, ε, συγγνώμη, για την Νότια Αφρική ε, παίξαμε το χαρτί αυτό και το κερδίσαμε. Για τη Δυτική Αφρική τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Εν πάση περιπτώσει αυτό που κάνω είναι ότι ακούω ό,τι έχουν να πούν τα, τα συνδικάτα, ακούω αυτές τις ιστορίες για τα παιδιά τα οποία δουλεύουν στη, στο κακάο και πραγματικά συγκινούμε κι εγώ γιατί άνθρωπος είμαι. Κοιτάξτε, τα χρήματα ε, δεν είναι το κεντρικό ζήτημα όταν ε, συζητάμε ε, για τα Economic Partnership Agreements. Είναι πολύ περισσότερο Αυτές οι EPA αφορούν πολύ περισσότερα πράγματα ε, και το ότι, ε, ε, το ότι αναγκαστήκαμε να δεχτούμε την ρήτρα μη εφαρμογή όταν αναγκάστηκα να τη δεχτώ ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα βλέπουμε ότι η κατάσταση μερικές φορές αλλάζει, ε, πρέπει να περιμένουμε λίγο μέχρι να ε, προχωρήσει η διαδικασία. Βλέπω ας πούμε τα νησιά του Σολομώντα τα οποία ε, έχουν κάποια προβλήματα. Δεν είναι, δεν είναι ψευτοσυμφωνία, μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένη, αλλά πάντως ε, είναι συμφωνία και έχω και την αίσθηση ότι ε, ο κόσμος, οι συμμετέχοντες ε, σκέφτονται πολύ περισσότερο και πολύ πιο συνολικά τα ζητήματα. Ενδεχομένως θα πρέπει να ανοίξουμε κάποια κεφάλαια όσον αφορά κυρίως την αηφόρο αλία που είναι πάρα πολύ σημαντική για τις περιοχές. Θα σας ενημερώνω και από την άλλη πλευρά, όπως κάνω και για πολλές άλλες περιοχές, εγώ προσπαθώ να βάλω στο παιχνίδι και την ε, ε ρήτρα της ε, αηφορίας. Ε, προσπαθούμε να οικοδομήσουμε και εμπιστοσύνη και προσπαθούμε και να περάσουμε τις πραγματικές αξίες τις οποίες έχει να δώσει η Ευρώπη. Όσον αφορά λοιπόν ε, τα συνδικάτα, όσον αφορά ε, τις, τις συνθήκες εργασίας, ναι, του συναντώ και, και, από την άλλη πλευρά να μην ξεχνούμε ότι οι κυβερνήσεις δεν δίνουν τα κείμενα στις, στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ή των ε, ε, συνδικάτων. Ε, συζητούμε βέβαια και είμαστε σε διαρκή επαφή και με τον Επίτροπο Σιόλος και φυσικά όλοι χαρήκαμε με τις γεωγραφικές ενδείξεις. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Τώρα, αυτό το θέμα της Αφρικανικής Ένωσης και του προβληματισμού για την ειλικρίνεια των προθέσεων. Δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς τα προβλήματα. Ε, πάντως εμείς, μπορούμε να εμείς αυτό που κάνουμε είναι ε, να προσφέρουμε καλές εταιρικέ συμφωνίες <clears throat> με τις χώρες ε, χωρίς ε, ε, κρυφά κεφάλαια και χωρίς φυσικά να αφαιρούμε τα προτιμησιακά καθεστώτα γιατί τα αντικαθιστούμε με άλλου είδους προτιμήσεις και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι με όλες τις χώρες του κόσμου και να έχουμε μια ίδια προσέγγιση. Τώρα, δεν είμαι βεβαία τι σημαίνει και τι ακριβώς αντιπροσωπεύει η έκφραση καλή την πίστη σε αυτές ε, τις ε, διαπραγματεύσεις. Ε, εμείς σίγουρα δεν έχουμε κρυφή ατζέντα. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία σίγουρα δεν είναι ιδεώδη, ίσως θα μπορούσαν να προωθηθούν με λίγο διαφορετικό τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει περιπτώσει προσπαθούμε να φτάσουμε, να επιτύχουμε ε, ε, ε, πράγματα τα οποία στην ουσία εκπροσωπούν και τις αξίες μας. Ε, απ' την άλλη πλευρά ε, είναι αλήθεια ότι ε, απέναντί μου έχω συχνά ανθρώπους που βλέπουν αυτές τις συμφωνίες ε, και με πολύ πατερναλιστικό τρόπο εμείς έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία και ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε, ε, που αφορούν την Συμφωνία για τη Δυτική Αφρική και που τα έχουμε αντιγράψει στην ουσία. Είναι αντιγραφή και επικόλυση του άρθρου 96 και κάποιων στοιχείων της Συμφωνίας του Κοτονού. Ε, ξέρετε ότι υπάρχουν ωστόσο κάποια στοιχεία που τους φοβίζουν ε, και νομίζω ότι η διέξοδος είναι μόνο η συζήτηση και όχι η ε, υποχρέωση να δεχτούν σκληρούς κανόνες. Ε, ερώτηση για αυτό το EAC για την Ανατολική Αφρική. Ναι, αναφερθήκατε σε αυτή τη ρήτρα του Most Favored Nation Μπορώ να σας δείξω και τα κείμενα αν θέλετε. Μπορώ, θα δείτε ότι δείξαμε πάρα πολύ μεγάλη ε, ευελιξία. Αυτή η περιφέρεια, ε, η, περιφέρεια της Αφρικής EAC ε είναι περίπλοκη. Δεν λέω, δεν θέλω να πω ότι η Νότια Αφρική είναι τελείως διαφορετική, αλλά de facto είναι διαφορετική η περιφέρεια EAC ε, όπως και σε άλλες ε, περιοχές ε, έχουμε άλλου είδους κατάσταση όσον αφορά τους δασμούς, τους εξαγωγικούς δασμούς και με κάποιο τρόπο θα πρέπει όταν αφαιρούμε εξαγωγικούς δασμούς να βάλουμε κάτι άλλο στη θέση τους και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις ε, τα προβλήματα είναι ε, ε, οικονομικά γιατί δεν καταφέρνουν ούτε καν να καλύψουν και τα έσοδα που χρειάζονται μέσα από αυτούς τους δασμούς και επομένως μερικές φορές πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο εύκολα τα κείμενα για αυτές τις περιοχές της ε, Αφρικής. Όπως σας έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, το μεγάλο πρόβλημα ε, για αυτή την περιφέρεια τουλάχιστον ε, για μία χώρα είναι η ρήτρα μη εκτέλεσης και το ζήτημα των, του MFN, Most Favored Nation και των εξαγωγικών δασμών δεν τα συζητήσαμε καν την τελευταία φορά. Δεν νομίζω ότι μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Ε, δεν, μπορώ να, δεν μπορώ να σας εξηγήσω και φυσικά δεν μας αρέσει αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με αυτή τη χώρα. Όσον αφορά τα Φίτζι, ναι, το 2006 πήραμε αυτή την απόφαση που αναφέρατε. Είναι γεγονός ότι τα Φίτζι όπως και η Μαδαγασκάρη ε, υφίστανται αυτές τις ε, κυρώσεις οι οποίες έχουν αρθεί τώρα για την περίπτωση των Φίτζι. Όσον αφορά την άναρχη αλληλεία και τα λοιπά, την IUU, ξέρουμε ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Ε, όταν ε, ε, έχοντας έρθει σε επαφή συχνά με τις χώρες αυτές πραγματικά αισθάνονται πολύ καλύτερα όταν βλέπουν ότι τους φερόμαστε σαν να είναι ισότιμοι συνομιλητές και πραγματικά νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε τίποτα τουλάχιστον δεν θα καταφέρουμε κάτι περισσότερο εάν κλείσουμε την πόρτα του στα νησιά αυτά και στις χώρες χώρες αυτές. Υπάρχουν χώρες όπως και η Σρι με την οποία γνωρίζω από πρώτο χέρι. Ε, ε ξέρω ότι εκεί δεν ε, κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά δεν μπορώ να πω ότι είμαι ε, περήφανη ε, ίσως, ίσως δεν είναι καθόλου ιδεώδης η κατάσταση αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθήσαμε έστω και με αυτή την από την πίσω πόρτα της κοινωνίας των πολιτών να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε κάποιες ανάγκες Uh, Έτσι πιέσαμε έμεσα την κυβέρνηση αυτών των χωρών και δεν θεωρώ ότι κάναμε λάθος. Μία ενδιαφέρουσα ερώτηση γιατί οι χώρες ΕΚΟΑΣΚ δεν έχουν ακόμη μονογράψει. Η κατεξοδότηση πράξης συγγνώμη, ναι, η κατεξοδότηση πράξης για την Ιγυρία και ίσως και για άλλες δεν υπήρχαν και εγώ δεν μπορώ να τις γεννήσω. Είναι θέμα διαδικασίες. Εμείς μορφωθήκαμε με τον νόμο και ελπίζω σε μερικούς μήνες ότι θα λυθεί το θέμα στις τρεις περιπτώσεις, ότι θα έχουμε υπογραφή μέχρι τέλους του χρόνου και μετά έχουμε τη διαδικασία επικύρωσης. Θα ωφελήσει όλες αυτές τις χώρες, γιατί θα έχουν το ίδιο καθεστώς. Χρειάστηκε να αποδεχθούμε ότι όλοι πρέπει να υπογράψουν, αλλά η επικύρωση πρέπει να είναι μόνο από τα τρία τέταρτα όπως το κοτονού και κατόπιν μπορεί να αρχίσει να ισχύει η συμφωνία για τις χώρες που την έχουν επικυρώσει. Εξαιρέθηκαν κάποιες χώρες. Θεωρείται ότι μπορούν να εξαιρεθούν, να μην επικυρώσουν δηλαδή. Ελπίζω όμως να επικυρώσουν όλες. Ελπίζω λοιπόν να λήξει αυτή η τρέχουσα κατάσταση που έχει να κάνει με τη φύση των συμφωνιών που είναι διαφορετικές. Χαίρομαι πάντα αντιμετωπίζω με ανάμεικτα συναισθήματα αυτές τις συμφωνίες. Κάποιες χώρες, όπως οι λιγότερο αναπτυξμένες χώρες, καταλαβαίνουν τι τους προσφέρει μια EPA. Αν έχεις μια τέτοια συμφωνία, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, αλλά η ουσία είναι, είναι ότι πολύ απλό να βοηθηθείς. Ενώ αν δεν έχεις μια τέτοια συμφωνία, είναι πολύ πιο περίπλοκο το καθεστώς. Είναι καλή περίπτωση για μια χώρα όπως σε Σενεγάλη να έχουν ΙΠΑ γιατί μπορούν να πυροδοτήσουν την τελευταία ρήτρα διαφύλαξης, να ενεργοποιήσουν την τελευταία ρήτρα διαφύλαξης την οποία τους παραχωρήσαμε και πρέπει να είμαστε περήφανοι. Ελπίζω να υπάρχει συνέπεια σε όλες μας τις ενέργειες αλλά βέβαια πάντα είναι καλοδεχούμενες συμβουλές για βελτίωση. Η ΑΕΤ μπορεί να επικυρώσει ή όχι αλλά είναι κρίμα που δεν επικυρώνουν γιατί είναι στο ίδιο νησί με το Δομήνικο. Και η EPA θα επέτρεπε να βελτιωθούν πολύ οι σχέσεις μεταξύ τους. Θα ήταν ένα περιφερειακό πλαίσιο, αλλά είναι δική τους η επιλογή. Α, η μελέτη για τις EPA, για την Καραϊβική, η μελέτη αυτή, την έχουμε. θα δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες μάλλον. Πρέπει να μας στείλουν ε, οι συντάκτες το τελικό κείμενο, δεν το έχουμε δει ακόμη. Μόλις μας τη στείλουν την τελική εκδοχή, με το τιμολόγιο θα τη βάλουμε στο site. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Κλείνουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ άλλη μια φορά. Περνάμε στο πρώτο τελευταίο, το 14. Ενημέρωση για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνία με το Εκουαδόρ για να συμπεριληφθεί στη συμφωνία που έχουμε εδώ και καιρό με την Κολομβία και το Περού. Αυτό ήδη αξίζει να το ακούσουμε, αλλά θέλουμε να μάθουμε τι θα γίνει με το Εκουαδόρ μέχρι να αρχίσει να ισχύει αυτή η επέκταση της συμφωνίας. Αυτή τη στιγμή έχουν ε, έχουν ε, καθεστώς γενικευμένων ε, προτιμήσεων συν και πρέπει να το συζητήσουμε. Ο κύριος Γιώργενσεν που τον έχουμε δει πολλές φορές να του δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει την ε, κατάσταση πραγμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσω για το πώς έχουν τα πράγματα στη διαδικασία αυτή με το Εκουαδόρ. Σημαντικές εξελίξεις είχαμε στο τέλος του καλοκαιριού και καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών εργαστήκαμε και τώρα εργαζόμεθα για να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο θέμα τι πρέπει να συμβεί μεταξύ της κατάληξης των διαπραγματεύσεων και της αρχής ισχύω για να μην υπάρξουν κολλήματα στο εμπόριο. Αλλά επειδή έχει περάσει καιρός από τότε που συζητήσαμε αυτό το θέμα τελευταία φορά, να σας ενημερώσω για το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και τη συμφωνία και μετά να δούμε ποια είναι τα ωφέλη γιατί είναι σημαντική συμφωνία και κάποια θέματα για το πώς και σε τι βαθμό μοιάζει ή διαφέρει αυτή η συμφωνία με τη συμφωνία που έχουμε με την Κολομβία και το Περού. Πρώτον λοιπόν, το ιστορικό. Η διαπραγματεύση ξεκίνησε το 2007 με τέσσερις χώρες για να καταλήξουν σε συμφωνία. Αυτή η διαδικασία ήταν δύσκολη. Υπήρχαν διαφορές προσέγγισης μεταξύ των χωρών αυτών και στην πορεία η Βολιβία αποφάσισε να αποχωρήσει. Οι άλλες τρεις χώρες, Εκουαδόρ, Περού και Κολομβία, συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις. Το Εκουαδόρ συνάντησε, ε, αποφάσισε να αναστείλει τη συμμετοχή του το 2009. Καταλήξαμε αυτό που αποκαλούμε η πολυμερή συμφωνία με την Κολομβία και το Περού τον Μάρτιο του 10. Η συμφωνία με το Περού και την Κολομβία άρχισε να ισχύει πέρυσι και από τη στιγμή αναστολή των διαπραγματεύσεων και σε όλη τη διαδικασία επικύρωση τη συμφωνία με το Περού και Κολομβία διατηρήσαμε επαφέ με το Εκουαδόρ για να του ενημερώνουμε. Και είχαν τη δυνατότητα να μελετήσουν αναλυτικά τη συμφωνία. Αυτή η διαδικασία κατέληξε, κορυφώθηκε μπορούμε να πούμε, σε μια υπουργικού επίπεδου συνάντηση πέρυσι τον Ιούλιο. Οπότε ξεκίνησαν ε, τεχνικές συναντήσεις και υπήρξε και μια συνάντηση με τον Επίτροπο και όλα αυτά επέτρεψαν να, να υπάρξει απόφαση να ξαναξεκινήσουν οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης με το Εκουαδόρ. Θεώρησαν ότι είναι καλή για αυτούς η κατάσταση και ότι αυτό που αποφασίσαμε με τον Περού και την Κολομβία μπορούσε να γίνει αποδεκτό και από εκείνους. Πήγε πολύ γρήγορα κατόπιν διαπραγμάτευση. Είχαμε μια ανταλλαγή προσφορών πριν το τέλος του χρόνου, 13, πρώτος γύρος τον Ιανουάριο, εδώ στις Βρυξέλλες, δεύτερος γύρος στο Εκουαδόρ, τρίτος γύρος στις Βρυξέλλες, οπότε και συμφωνήσαμε τον Ιούνιο επί των περισσότερων θεμάτων οι δύο πρώτοι γύροι ήταν προπαρασκευαστικοί. Στον τρίτο γύρο είχαμε ουσιώδη πρόοδο. Μόνο λίγα θέματα έμειναν. Και στον τέταρτο γύρο τον Ιούλιο στις Βρυξέλλες που σε λίγο πάνω από δύο εβδομάδες καταλήξαμε σε τελική συμφωνία για όλα τα εκκρεμούντα θέματα Και είχαμε και μια συνάντηση τελική σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του Επιτρόπου Ντεχούκτου και του Εκουαδοριανού Υπουργού Εμπορίου. Υπήρξε λοιπόν πολιτική κατάληξη τον Ιούλιο, πριν από δύο μήνες. Και τώρα κάνουμε τον νομικό έλεγχο του κειμένου είναι προσχώρηση σε υπάρχουσα συμφωνία. Οι αλλαγές ε, είναι περιορισμένες. Εάν είστε επιμελής, εμπορικών, επιμελής, επιμελής μελετητής εμπορικών συμφωνιών, μπορείτε να τις μελετήσετε. Είναι στο διαδίκτυο για λόγους διαφάνειας. και για να ενημερώσουμε τους εταίρους μας. Χθες μπήκε στο διαδίκτυο φρέσκο. Έχει δύο τμήματα. Ένα, αλλαγές στο κείμενο της συμφωνίας και τα χρονοδιαγράμματα πρόσβασης στις αγορές για το Εκουαδόρ και για μας και αν δείτε το κείμενο είναι πολύ περιορισμένες οι αλλαγές. Έχουμε τρία είδη τροποποίησεων. Πρώτο είδος, οι αναγκαίες αναφορές στο Εκουαδόρ και τις αρχές του, Βεβαίω έχει αλλάξει και το άρθρο που αναφέρεται στις περιοχές που καλύπτει η συμφωνία. Κατόπιν σε 12 σημεία προσαρμόσαμε το κείμενο για να δούμε τις διαφοροποιήσεις των δεσμεύσεων του Εκουαδόρ. Αυτή η διαφορετικότητα της αντιμετώπισης προβλέπεται και για την Κολομβία και το Περού, για παράδειγμα, για τις υπηρεσίες, όπου υπάρχει ο ορισμός της εθνικής αντιμετώπισης. Και ένας κατάλογος τομέων, στον τομέα των υπηρεσιών που υπάρχει χωριστή αντιμετώπιση και μια τελική ομάδα προσαρμογών του κειμένου που είναι ειδικέ υποσημειώσεις που αναφέρονται στην ειδική μεταχείριση που χρειάζεται το Εκουαδόρ λόγω ειδικών καταστάσεων που ε, προκύπτουν από το συντάγμα τους, από το νομικό τους πλαίσιο ή για άλλους πολιτικούς λόγους. Για παράδειγμα, επιθυμούσε το Εκουαδόρ να έχει την δυνατότητα στην ε, Εμπορική Επιτροπή να δει τι επιπτώσεις θα έχει η συμφωνία στις λεγόμενες ενώσεις ε, αλληλέγγυας και λαϊκής κατανάλωσης που είναι ενώσεις που υπάρχουν για να βοηθήσουν την ανάπτυξη της, ε, εκουαδοριανής κοινωνίας. θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές περιορισμένες και έγιναν για λόγους σωστής νομικής τάξης και για να λάβουν υπόψη τις πολιτικές ευαισθησίες και τις ανάγκες που προέβαλε το Εκουαδόρ. Σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά ε, και τις δεσμεύσεις, ε, σχετικά με το Εκαδόρ, όλα τα έχετε, είναι γραμμένα. Ε, ε, βέβαια το κείμενο ακόμα δεν το έχουμε, δεν έχει ελεγχθεί νομικά. Ε, εν πάση περιπτώσει όμως ε, υπάρχουν πολλά συγκρίσιμα σημεία ε, και τουλάχιστον σε ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας με αυτά που είχαμε συμφωνήσει με το Περού και την Κολομβία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Ε, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά στις υπηρεσίες. Ε, εκεί το Περού και η Κολομβία δεν άνοιξαν τα κεφάλαια, ούτε και το, ούτε το άλλωστε. Υπάρχουν όμως άλλα κεφάλαια ε, τα οποία έχει ανοίξει το Εκουαδόρα ενώ δεν έχει πράξει ομοίως η Κολομβία, ούτε όμως και το Περού. Ε, κίνηση ε, ατόμων, ελεύθερη κυκλοφορία. Ε, Ιδίω δεν λαμβάνονται υπόψη τα αιτήματα τα εξειδικευμένα της χώρας. Όσον αφορά τα αγαθά, είναι μια καλή συμφωνία το Εκουαδόρ στο τέλος της απόφασης ε, θα ε, απελευθερώσει 97% της ε, αγοράς περίπου για 10 χρόνια για τα περισσότερα αγαθά ε, θα υπάρξει μια περίοδος μεταβατική με ένα ποσοστό περίπου 60%. Επίσης θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και για κάποια εξαιρετικά ευαίσθητα προϊόντα για το Εκουαδόρ. Και εν θα καλέψουμε περίπου 99,6% όλων των ε, τρέχουσών εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα. Αυτό ε, είναι απολύτω συγκρίσιμο με τα επιτεύγματα των αντιστοίχων συμφωνιών με την Κολομβία ε, και το Περού, γιατί και εκεί είμαστε περίπου στα ίδια ποσοστά. Οι υπηρεσίες τώρα, και εδώ είναι εξισορροπημένη η συμφωνία, Εξίσου φιλόδοξο το πρόγραμμά μας με την Κολομβία και το Περού και απλώς παραμένουν θερματοπιστωτικές υπηρεσίες, ε, ε, τηλεπικοινωνίες, ε, υπηρεσίες διανομής κλπ. Δημόσιες προμήθειες τέλος. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό σημείο για μας. Το Εκουαδόρο συμφώνησε να ανοίξει τις αγορές του στο ίδιο επίπεδο με την Κολομβία και το Περού. Υπάρχουν κάποιες διαφορές εδώ, οι οποίες οφείλονται ε, στο ότι όταν ε, κάποιος διαπραγματεύεται μια συμφωνία και όταν ας πούμε ανοίγει το κεφάλαιο για τις ε, προμήθειες δεν είναι πλήρες το άνοιγμα, δηλαδή υπάρχει πάντα η δυνατότητα της χώρας να πει δεν θέλω να ανοίξω ακριβώς αυτό τον τομέα, μπορώ όμως να ανοίξω περισσότερο έναν άλλον, υπάρχουν κάποιες διαφορές πάντα ναι, και στην προκειμένη περίπτωση του Εκουαδόρ υπάρχουν κάποιες διαφορές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες, συμφωνίε συμφωνίες με την Κολομβία και το Περού. Λάβαμε υπόψη σε αυτό το τμήμα το χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης συγκρίνοντας το Εκουαδόρ με την Κολομβία και το ε, Περού, ε, βλέπετε τη διαφορά αυτή και αυτή η διαφορά ελήφθη υπόψη εν είδη μεταβατικών περιόδων στο Εκουαδόρ, ας πούμε όσον αφορά τα κατόφλια ε, σχετικά με το πότε θα πρέπει να ανοίξουν οι δημόσιες προμήθειες και οι αγορές τους. Τα επόμενα βήματα. Τώρα έχουμε ξεκινήσει την διαδικασία της νομικής αναθεώρησης Παίρνει λίγο χρόνο, αλλά έχουμε καλή, καλό ρυθμό και ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε την ε, νομική αναθεώρηση μέχρι τον Νοέμβριο. και σε αυτήν την ε, διαδικασία βεβαίως να ολοκληρώσουμε και το πρωτόκολλο ε, ένταξης. Προσχώρηση, συγγνώμη, και το πρωτόκολλο προσχώρησης, ε, όπως κάναμε ακριβώς και με την Κολομβία και το Περού γιατί βεβαίως για να τεθεί σε ισχύ ε, η συμφωνία αυτή θα πρέπει να ε, συμφωνηθεί και από την αντίστοιχη επιτροπή που είναι βεβαίως το υψηλότερο σώμα ε, της επαφής που έχουμε με την Κολομβία και το Περού και εκεί η Κολομβία και το Περού έχουν δυνατότητα ανασχετικής ψήφου. Τώρα, το πρωτόκολλο θα πρέπει να εγκριθεί από την ε, Επιτροπή που αποτελείται από τις χώρες αυτές και οι σχετικές προτάσεις θα για ε, υπογραφή θα ε, διαβιβαστούν στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σε ένα χρόνο περίπου από τώρα, γύρω στον Οκτώβριο του 2015. Ε, θα έχουμε λοιπόν υπογραφή και επομένως ε, και πρώτη μεταβατική εφαρμογή υλοποίηση αρχές του 2016. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπατε κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά ε, το θέμα των γενικευμένων προετοιμήσεων. Η κατάσταση είναι η εξή. Το Εκουατόρ θα χάσει την, ε, ε, το, το GSP Plus μέχρι το τέλος του χρόνου, αυτό είναι αναπόφευκτο. Ωστόσο, είναι εξίσου σαφές ότι τώρα η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι διαφορετική. Δηλαδή έχει ολοκληρωθεί μια εμπορική συμφωνία με το Εκουαδόρ. Έχουμε φτάσει στην πολιτική ε, ε, ολοκλήρωση της συμφωνίας και προχωρούμε με τα ε, τεχνικά στοιχεία τα οποία θα ολοκληρώσουν την πρόταση και με την νομική αναθεώρηση. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για μια προτιμησιακή σχέση όσον αφορά το ε, εμπόριο. Αυτό σημαίνει ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Εκουαδόρ θα κάνουν προσπάθεια έτσι ώστε να γεφυρώσουν το χάσμα ε, ανάμεσα ε, στην εκπνοή του συστήματος GSP και την εφαρμογή της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου. Ε, ε, ε, στο εσωτερικό της υπηρεσίας δουλεύουμε για να δούμε, να βρούμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα έχει σκαμπανεβάσματα. ε, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη κάποια ιδιαίτερα εξαγωγικά κεφάλαια για το Εκουαδόρ. Ε, και εδώ μιλάμε για αύξηση των ε, δασμών της τάξης περίπου του 24% που μπορεί να έχει πολύ μεγάλη επίπτωση σε την ροή των εξαγωγών και την εισαγωγή προϊόντων του Εκοδόρου στην αγορά μας. Η ιδέα μας λοιπόν θα ήταν θεωρητικός Η ιδέα μας λοιπόν θα ήταν ε, να προετοιμαστούμε καλά για αυτήν την ε, συμφωνία ε, έχοντας ένα αμοιβαίο stand still. Μία παύση δηλαδή, στη διάρκεια της οποίας δεν θα εισαχθούν νέα μέτρα, δεν θα αυξηθούν οι δασμοί ή δεν θα υπάρξουν άλλου είδους περιορισμοί. Αυτή είναι η γενική ιδέα. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στην προετοιμασία του όλου ζητήματος και ευελπιστούμε ότι θα είμαστε σε θέση να στείλουμε την πρόταση της Κομισιόν ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές Οκτωβρίου και βεβαίως ε, μιλώ υπό την αίρεση των αποφάσεων ε, του κολεγίου που θα πρέπει, το, που θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, εγκρίνει την πρόταση ή βρίσκεται στην ημέρηση, θα βρίσκεται στη μεσή διαταξή τους αρκετά σύντομα. Έχουμε προχωρήσει, χρειαζόμαστε όμως και την τυπική επικύρωση. Τελειώνω, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, μην ανησυχείτε προχωρήσαμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά πρέπει να σας πω ότι τον Ιούλιο ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και δεν είχαμε ε, την δυνατότητα να σας πούμε οτιδήποτε πριν από το πέρας των διαπραγματεύσεων. Έχουμε 10 λεπτά, λέει ο Πρόεδρος ακόμα. Γι' αυτό όσοι θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις, παρακαλώ ε, ε, σύντομα. Έχουμε τον μόνιμο εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την αναλυτική παρουσίαση και για το πόσο επιχείρηση να είναι διαφανής όσον αφορά τη διαδικασία για το πώς προέκυψε αυτή η Συμφωνία Ελευθερομπορίου. Τον Απρίλιο, συγγνώμη την Άνοιξη, είχαμε διάφορες συναντήσεις της ομάδας ε, παρακολούθησης της συμφωνίας ε, για το Περού και την Κολομβία και θα κάνουμε προσεχώς και άλλες τέτοιες συναντήσεις για να δούμε τι θα γίνει τώρα με την προσχώρηση και το Εκουαδόρ. Αλλά πρέπει να μπει σε ένα γενικό πλαίσιο και κατά τη γνώμη μου ως Επιτροπή πρέπει να καλύψουμε δύο προκλήσεις εγκαίρως. Είπατε ότι τι θα γίνει από πρώτης πρώτου. Εάν δεν έχουμε βρει λύση, θα καταργηθεί το καθεστώς γενικευμένων προτιμήσεων για το Εκουαδόρ Βέβαια είναι σύντομο το διάστημα για να εγκρίνει η Κομισιόν ένα τέτοιο κανονισμό. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε στο Εκουαδόρ όλες τις δυνατότητες που έχουν αυτή τη στιγμή πρόσβαση στην αγορά της Ένωσης. Παρακαλώ την Κομισιόν έγκαιρα να μας στείλει πρόταση κειμένου για να μπορέσουμε μέσω της ε, τακτικής νομοθετικής διαδικασίας να το, να το εξετάσουμε. Πρέπει να το ελέγξουμε. Δεν είμαστε απλώς για να εγκρίνουμε όπως συνέβη με κάποια άλλα επίγοντα θέματα. Θέλω να αποφύγω τέτοιες καταστάσεις. Και δεν θέλω να διακινδυνεύσουν οι διμερείς μας σχέσεις. Δεύτερον, είχαμε επιμείνει ως κοινοβούλιο σε έναν οδικό χάρτη που να συνοδεύει την ε, σύμβαση με το Περού και την Κολομβία. Θέλουμε λοιπόν και τώρα έναν οδικό χάρτη που να λαμβάνει υπόψη όλες τις ε, επιπτώσεις της ε, προσχώρησης του Εκουαδόρ. Και ίσως θα πρέπει να υπάρχει και ένα συνοδευτικό ψήφισμα ακόμη και για αυτό το πρώτο τμήμα πριν εγκρίνουμε τη συμφωνία που να αναφέρει τις ε, κοινωνικές πολιτικές του Εκουαδόρα για να δώσουμε στη χώρα μια δυνατότητα να καταλάβει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί και υποστηρίζουμε αυτή την πορεία της κυβέρνησης και της κοινωνίας στο Εκουαδόρα. Και θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν όλες τις οικολογικές προκλήσεις που αναφέρονταν και στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου όταν συζητήσαμε όταν συζητήσαμε το ψήφισμα για τις σχέσεις, μας, τις σχέσεις μας με τη Λατινική Αμερική. Και τέταρτον, θέλω να συνεργαστούμε στενά με όλους τους σκιώδεις. Θα καλωσόριζα λοιπόν ορισμό σκιωδών από όλες τις ομάδες και θέλω να ε, Έχω και τη βοήθεια της γραμματείας. Ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ πρόεδρε και γρήγορα να σας πω. Χαίρομαι που ολοκληρώσαμε αυτές τις συνομιλίες με το Εκουεδόρ και ξεπερνώντας ορισμένες διαφορές ιδεολογικές, ε, ίσως η Βολιβία δεν τις ξεπέρασε αυτές. Η συμφωνία θα μπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα, αποδειχθεί ιδιαίτερα θετική και σχετικά με την Ισπανία και τα Κανάρια νησιά ίσως υπάρξει ένα κάποιο προβληματάκι σχετικά με τις μπανάνες αλλά σε παρόμοιες συμφωνίες τι να κάνουμε ε, κάτι όλο και κάτι εμφανίζεται ιδιαίτερα σημαντικό νομίζω ότι στο χρονικό αυτό διάστημα από τη στιγμή της λήξεως ε, της σημερινής συμφωνίας ε, Συν ε, όταν θα ισχύσει αυτή η συμφωνία με το Εκουαδόρ και η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει κάτι γιατί φαίνεται καθαρά εδώ ότι διαφορετικά θα έχανε ιδιαίτερα το Εκουαδόρ στην περίπτωση αυτή. Πάντως είμαι στη διάθεσή σας, είμαι από το ΕΛΚΟΣ και ο και για παρόμοια ε, θέματα, για παρόμοιο τύπου διαπραγματεύσεις. Um, um, come back Ευχαριστώ. Αυτό που είπε ο θέλω και εγώ να αναφέρω για τον οδικό χάρτη δεν είναι μόνο ένας οδικός χάρτης αλλά και το κεφάλαιο της συμφωνίας για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι το Εκουαδόρ έχει γίνει αντικείμενο συστάσεων από το Γραφείο Εργασίας επανειλημμένα συγκεκριμένα γιατί δεν συμμορφούνται με τις αποφάσεις του ILO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την ε, ελευθερία του συνεταιρίζεστε και τις ελεύθερες λογικές συμβάσεις. Ξέρω επίσης ότι λαμβάνουμε όλο και περισσότερη πληροφόρηση από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και από τις συμβουλευτικές επιτροπές του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της συμφωνίας με την Κολομβία και το Περού. Θα καλούσα το Χέλμουντ να υπάρξει απόφαση εντός της Επιτροπής μας, αλλά να την επεκτείνουμε για να εξετάσουμε πώς λειτουργεί ο δικός χάρτης για τις τρεις χώρες και πώς λειτουργούν οι ε, εθνικές επιτροπές ε, παρακολούθησης του κεφαλαίου για την βιώσιμη ανάπτυξη γιατί όλες μας οι πληροφορίε είναι ότι υπάρχουν προβλήματα και χθε λυπήθηκα πολύ που άκουσα ότι δολοφονήθηκαν στην Κολομβία άλλοι δύο συνδικαλιστές πρέπει πολλά να κάνουμε και πρέπει το Εκουαδόρ να προσχωρήσει σε ένα σύστημα που να λειτουργεί και όχι που δεν λειτουργεί όπως και ζούνται αν δεν κάνω λάθος και ρωτάω την Επιτροπή η συμφωνία με την Κολομβία δεν έχει επικυρωθεί από όλε τι χώρε, αν δεν κάνω λάθο. Το Βέλγιο είναι από τι χώρε που δεν επικύρωσε ακόμα τη συμφωνία με την Κολομβία. Ίσως δημιουργήσει πρόβλημα και σήμερα στην Κολομβία. Γιατί? Το, ενώ το συνταγματικό δικαστήριο φρονεί ότι αυτή η συμφωνία δεν ε, είναι αντισταγματική. λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Μήπως υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα μήπως θα πρέπει να αφαιρεθούν αυτοί οι λόγοι και το είπαμε προηγουμένως για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, την προστασία των μειονοτήτων και του περιβάλλοντος στα θέματα που είχαν τεθεί κανονικά συμφωνία με την Κολομβία. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε κάτι σαν εργασία για να μπορέσει να επικυρωθεί παντού αυτή η συμφωνία από τα κράτη-μέλη και να ξεφύγουμε από τη σημερινή κατάσταση σχετικά με τη συμφωνία με την Κολομβία και να συμμετάσχουν όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σάντσες. Ακόμα μια φορά, να που είμαστε θεατές και συνένοχοι, δεν είναι τόσο εμπορική, είναι γεωπολιτική συμφωνία, οικονομική και με περιφερειακή εναλλακτική λύση στην περιοχή. Αυτά είναι άδικα, άδικα, γιατί δεν υπάρχει συμμετρία ανάμεσα στα δύο μέρη. Αυτό φαίνεται καθαρά. Εδώ θα είναι απεικιοκρατική υπέρ της εξορρεκτικής βιομηχανίας και πρωτογενών προϊόντων έτσι, που ε, είναι των μεγάλων εταιριών των ευρωπαϊκών κυρίως και του Εκουαδόρ ακόμα και θα έχουν έτσι επιπτώσεις ε, περιβαλλοντικές κλπ που δεν ελήφθησαν υπόψη στις ε, διαπραγματεύσεις και επίσης ε, και τα κράτη δεν μπορούν να επέμβουν οικονομικά, επίσης στα τρόφιμα, στην εξασφάλιση τροφίμων και στα ε, εργασιακά και στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κολομβία. Αυτά λοιπόν, όπως είπε και ένα προηγουμένως, ε, Αυτά είναι μου. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το ανθρώπινο είδος. Η Επιτροπή τι κάνει μετά από την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου, του συνταγματικού δικαστηρίου που λέει ότι είναι αντισυνταγματικός αυτός ο νόμος. Ε, εντάξει και για τη ρήτρα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι γίνεται, γιατί δεν διακόπτει, δεν παγώνει τη συμφωνία και να, πει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η ρήτρα από την Κολαβία. Και τελευταίο ελπίζουμε το ίδιο πράγμα όπως και με το Εκοδόν. Ναι, ένα λεπτό, ένα λεπτό εσύ. Έχω πολλές ερωτήσεις, οι οποίες όμως ε, δεν θα απαντηθούν γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο ε, για συζητήσεις. Ο κύριος Γιώργενσεν ε, πήρε όλο το χρόνο που είχαμε προβλέψει με την αρχική του παρέμβαση, πήρε όλο το χρόνο που είχαμε προβλέψει για αυτή την συζήτηση. Ήταν ένας μακρύς μονόλογος και τώρα δεν έχουμε την δυνατότητα. Δύο λεπτάκια έχουμε να μιλήσουμε ενώ θα έπρεπε να έχουμε 20. Άρα δεν μπορώ να υποβάλω πολλά ε, τα ερωτήματα μου όλα, μία μονάχα. Ε, ε, ε, έχουμε δυνατότητα σαν κράτη-μέλη να μην προσυπογράψουμε τη συμφωνία αυτή και να μου, κάνει, να μου δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση. Σήμερα είχαμε την πρώτη συζήτηση όπου είναι θέμα ενημέρωσης και φυσικά θα εμβαθύνουμε και δεύτερον θεωρώ ότι η ομάδα παρακολούθησης όταν οριστούν οι σκιώδεις θα συγκροτηθεί θα έχει περισσότερη δυνατότητα να συζητήσει. Κύριε Γιώργενσεν, τρία λεπτά. Τρία λεπτά για να απαντήσετε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα η φόρος ανάπτυξη είναι, είναι ε, τμήμα της ε, συμφωνίας την προσυπέγραψε, ε, προσυπέγραψε το τμήμα αυτό και ε, το Εκουαδόρ, το οποίο βεβαίως θα πρέπει να έχει τις ίδιες ε, υποχρεώσεις με το Περού και την Κολομβία. Και επίσης θα υπάρξει προσπάθεια επιθεώρησης και αναφοράς από τη δική μας πλευρά και που βεβαίως θα υποβάλουμε τις αναφορές μας στο Κοινοβούλιο όπως προβλέπεται και στον ε, αντίστοιχο κανονισμό ο οποίος ε, συνεφωνήθη μαζί, ε, ταυτόχρονα με, τον, με την διαπραγμάτευση για τη συμφωνία αυτή. Ένα χρόνο μετά την, το πρώτο έτος εφαρμογής ε, μάλλον υπογραφής, θα έχουμε ολοκληρώσει και τη μετάφραση κτλ. Και, ε, και ε, σας είπα ότι το Νοέμβριο θα στείλουμε από ό,τι φαίνεται κατά πάσα πιθανότητα την έκθεση στο Κοινοβούλιο. Και σας λέω ότι υπάρχει ιδιαίτερη υπογράμμιση του θέματος της αηφόρου ανάπτυξης. Είναι γεγονός ότι δεν έχει επικυρωθεί σε όλα τα κράτη-μέλη η συμφωνία αυτή από όλα τα κράτη-μέλη. Ε, συμφωνώ απολύτως με το Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει ε, να προσπαθήσουμε ε, να έχουμε πλήρη επικύρωση από όλες τις χώρες γιατί με τον τρόπο αυτό θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα πολιτικό προς το Περού και την Κολομβία ότι πρόκειται για μια συμφωνία την οποία λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και τη θεωρούμε σημαντική. Κυρία Κέλλερ, ναι, οπωσδήποτε τα κράτη-μέλη θα ε, εμπλακούν στην διαδικασία, θα συμφωνήσουν, θα επικυρώσουν μάλλον την συμφωνία ε, αυτή ίσως με τον, τρόπο, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ε, είχαν ενεργήσει για το Περού και την Κολομβία. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Θα κάνουμε ακριβώς τις ίδιες προτάσεις με αυτές που είχαμε κάνει για το Περού και την Κολομβία και θα ακολουθηθεί η ίδια νομοθετική διαδικασία όπως για το Περού και την Κολομβία. Υπήρξε ένα ερώτημα όσον αφορά ε, την ε, συνταγματική συμβατότητα. Το μόνο που μπορώ να πω για αυτό, για την κατάσταση που έχει προκύψει στην ε, Κολομβία, είναι ότι η παρούσα διαδικασία που είναι συνταγματική διαδικασία θα προχωρήσει η διαδικασία αυτή ε, και δεν προβλέπουμε να προκύψουν προβλήματα όσον αφορά την ίδια τη συμφωνία ή όσον αφορά τον σεβασμό της ε, ε, Κολομβίας στους όρους που εκεί προβλέπονται και την υλοποίησή τους. Βεβαίω είμαι στη διάθεση των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διμερώς να μου απευθύνουν ερωτήματα. Ευχαριστώ κύριε Γιούγκενσεν. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι στο θέμα της παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής των απαιτήσεών μας θα μας απασχολήσει και η Κομισιόν ίσως θα έπρεπε να προωθήσει αυτή τη διαδικασία ε, παρακολούθησης και θα το συζητήσουμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Διάφορα δεν υπάρχουν. Η επόμενη συνεδρίαση 6 και 7 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Η γραμματεία μου λέει είναι σημαντικό στις 29, 29 Σεπτεμβρίου ακρόαση των ε, νέων επιτρόπων. Ευχαριστώ πολύ.